Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα το απόγευμα, όπως βλέπετε, είμαστε αρκετά απασχολημένοι, το οποίο σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουμε το χρόνο μας. Θα δούμε την έκθεση Σαρακιάνη, όλοι θα έχετε το λόγο, χρειαζόμαστε αρκετό χρόνο δηλαδή, θα ήθελα όμως να είσαστε πειθαρχημένοι και να μας ε, πείτε αρκετά νωρίς κατά πόσο θέλετε το λόγο, έτσι ώστε να έχω τον κατάλογο και μετά να επιμερίσουμε το χρόνο ανάλογα με τον αριθμό των ομιλητών. Μετά από αυτή την έκκληση, την έκκληση θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Σαρακιάνη να λάβει το λόγο για τον, ε, σε σχέση με τον ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο. Έχετε το λόγο κυρία Σαρακιάνη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω για την εργασία και συνεργασία όλους τους σκιώδεις και τη γραμματεία της ΤΡΑΝ για την εργασία αυτή που ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη. Στόχος της αναδιατύπωσης είναι να φτάσουμε σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πρότυπο έτσι ώστε να έχουμε σαφείς κανόνες για να φτάσουμε σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο για να μην υπάρχουν επικρίσεις από το πρώτο, την εφαρμογή του πρώτου πακέτου. Εξού και η αναδιατύπωση. Στόχος λοιπόν είναι όχι να επιλέξουμε ένα από τα προϋπάρχοντα πρότυπα, αλλά ένα άλλο ενιαίο που να μπορεί να εφαρμοστεί από όλα τα κράτη-μέλη για να φτάσουμε στους βασικούς στόχους της ενιαίας αγοράς, καθώς και τους στόχους απομάκρυνσης των ε, ορυκτών καυσίμων, δηλαδή και την απομάκρυνση του διοξιδίου του άνθρακα και για να είναι το σύστημα αυτό ανταγωνιστικό. Οι βασικές πτυχές της ε, πολιτικής σειροδρόμων σχετίζονται με πέντε σημεία. Χρηματοδότηση, η αίρα, το διαχωρισμό μεταξύ υποδομών και αίρα, απελευθέρωση και εναρμόνιση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι όλες οι πτυχές ε, εντάσσονται σε αυτή την αναδιατύπωση. Ασχολήθηκαμε με τη χρηματοδότηση των σιδηροδρόμων και με τη ρυθμιστική αρχή και αποφάσισα το θέμα του unbundling, του διαχωρισμού, να το δούμε κατά μέρος. Δηλαδή, το 2000, με βάση το 2012, όπως μας είπε και, ο και η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της. Μιλάμε για μια αγορά που ήδη έχει απελευθερωθεί από το 2007 ε, για τα εμπορεύματα και από τον Ιανουάριο του 2010 όσον αφορά τους επιβάτες. Είμαι πεπισμένη ότι για το σιδηροδρομικό σχήμα χρειάζονται κανόνες και για τις πέντε αυτές πτυχές που δεν καλύπτει πλήρως το, η αναδιατύπωση και ένας ε, ρυθμιστής, ενιαίος ρυθμιστής, δεν μπορεί να καλύψει όλες τις πτυχές. Επίσης, ένα απελευθερωμένο σύστημα χωρίς το unbundling θα είναι ένα σύστημα που θα ενέχει διακρίσεις. Άρα χωρίς unbundling, χωρίς διαχωρισμό και απελευθέρωση δεν θα μπορέσει να ε, λειτουργήσει ένα σύστημα το οποίο θα πρέπει να έχει ίδια χρηματοδότηση. Γι' αυτό θα πρέπει να επέμβουμε και ως προς την τεχνική εναρμόνιση. Διαφορετικά δεν θα είναι δυνατόν να αναπτυχθεί ο τομέας. Άρα στο Recast θα ασχοληθώ με την ε, χρηματοδότηση, τη ρύθμιση και τον διαχωρισμό unbundling, όπως ορίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξεκινώ από ένα από τα βασικότερα σημεία της αναδιατύπωσης, δηλαδή του ε, ρυθμιστή. Τροπολογίες 73 μέχρι 88. Έτσι ώστε ο εθνικός ρυθμιστής να μπορέσει να λειτουργήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά μπορεί να μπορεί να προβεί και σε έναν σαφή διακανονισμό με βάση προγενέστερους κανονισμούς και έλεγχο της εφαρμογής των κανόνων στην αγορά των σιδηροδρόμων. Γι' αυτό έχω υποβάλει τροπολογίες για να είναι πιο σαφής η γνωμοδότηση. Δηλαδή, σε σχέση με την αδειοδότηση, τροπολογία 75 ή την οργανωτική υποδομή της τροπολογίας 73. Με απασχόλησε και το σκέλος της λήψης αποφάσεων, τροπολογία 80. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει καλύτερος έλεγχος και γι' αυτό ακριβώς μιλώ για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου ρυθμιστών που να είναι η βάση που να μπορεί να χρησιμοποιήσει ο ενιαίος Ευρωπαίος ρυθμιστής. Και επειδή δεν μπορεί να προβλεφθεί κάτι τέτοιο στο, στην αναδιατύπωση. Στην τροπολογία 88 ενέταξα αυτό το στοιχείο. Δηλαδή, μιλώ για το γεγονός ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί η αρχή του ενιαίου Ευρωπαίου ρυθμιστή. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα της χρηματοδότησης και του κόστους το γεγονός ότι είναι λίγες οι επενδύσεις στον τομέα των σιδηροδρόμων είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Δεν μπορεί να αναπτυχθεί ο τομέας όπως θα έπρεπε. Γι' αυτό θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σιδηροδρόμων να έχει τις κατάλληλες υποδομές για να είναι πιο ανταγωνιστικό πολλά κράτη-μέλη δεν έχουν λάβει επαρκώς υπόψη τη χρηματοδότηση των δικτύων, λαμβάνοντας υπόψη, μάλλον δίνοντας προτεραιότητα στις οδικές μεταφορές. Γι' αυτό υποστηρίζω την πρόταση της Επιτροπής έτσι ώστε να έχει ως πάγια διαδικασία τις πολιετής συμβάσεις στα κράτη-μέλη. Υπ' αυτή την έννοια θεώρησα ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τη διάρκεια της συμφωνίας από 5 σε 7 χρόνια για να υπάρχει καλύτερη αξιοπιστία του τομέα σε σχέση με τη διαμόρφωση του κόστους ως προς την αποδοτικότητα και την ηχορύπανση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το εξωτερικό κόστος και να το συντονίσουμε με άλλα μέσα μεταφοράς μέσα στα πλαίσια των διατροπικών μεταφορών. Γι' αυτό θεώρησα ότι θα πρέπει να συνδέσουμε τις σιδηροδρομικές μεταφορές με τις οδικές και να δώσουμε ένα μπόνους για να υπάρχουν επαρκείς επενδύσεις. Το σύστημα ε, λοιπόν των κινήτρων θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Διότι θα ήταν σκοπιμότερο να μην αλλάξουν οι υποδομές, αλλά να βελτιωθούν. Γι' αυτό δεν θα υπάρχει επιπρόσθετο κόστος, όπως προβλέπει η τροπολογία 62. Υπάρχει και ένα σύστημα bonus μάλους για να ενθαρρύνουμε για την χρήση, υπέρ της χρήσης των ε, τρένων και θεωρώ ότι οι υποδομές μπορούν να βελτιωθούν. Πιστεύω λοιπόν ότι με αυτό το σύστημα bonus μάλους θα ενθαρρύνουμε την χρήση των τρένων όπως ορίζει και η τροπολογία 76. Επίσης θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο κίνητρο για τη χρήση των τρένων όπως ορίζεται στην τροπολογία 127. Σε σχέση με τις κατεξουσιοδότηση πράξης Υπάρχουν 12 και μπορούν να αλλάξουν με βάση αυτό το μέσον. Θεώρησα λοιπόν ότι όλα αυτά θα είχαν επιπτώσει στο τελικό κείμενο της πρότασης οδηγίας. Γι' αυτό πρότεινα ορισμένες τροπολογίες έτσι ώστε τα παραρτήματα να ενταχθούν στην ομοθετική διαδικασία. Πρόκειται για τα παραρτήματα 2, 3, 4, 7 και 8. Άλλα τμήματα ίσως ορίζονται καλύτερα ως έχουν μέσα στα πλαίσια της εντολής. Επίσης, λαμβάνουμε υπόψη τις τροπολογίες δυνάμει της συνθήκης της Λισαβόνας με τις κατεξιοδότηση πράξης ως προς τις προβλέψεις της αναδιατύπωσης λαμβάνουμε υπόψη το unbundling, δηλαδή το διαχωρισμό μεταξύ φορέων και υποδομών. Μιλάμε για τις τροπολογίες από 17 μέχρι 28 και πιστεύω ότι αυτή η διάταξη θα πρέπει να ενταχθεί στην αναδιατύπωση. Πρότεινα λοιπόν έναν διαχωρισμό στο εσωτερικό του συστήματος των ε, σιδηροδρομικών μεταφορών και κατά την άποψή μου αυτό είναι ένα σωστό βήμα για να δούμε τι θα κάνουμε το 2012 με το άνοιγμα των αγορών, με την απελευθέρωση για να ανοίξουν οι αγορές. Πιστεύω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτό το πρότυπο. Διαφορετικά θα διευκολύνουμε μόνο τον ε, μεγάλο οικονομικό φορέα που κατέχει δεσπόζουσα θέση, έτσι κι αλλιώς. Έτσι δεν μπορούν να μπουν νέοι οικονομικοί φορείς, ιδιαίτερα από τις όμορες χώρες και αυτό θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις επί του ανταγωνισμού. Επίσης, αυτό αφορά την ανάπτυξη αγοράς και τους ε, διεθνικούς φορείς, διακρατικούς φορείς, επειδή μιλάμε για την απελευθέρωση των εμπορευμάτων και της ε, μεταφοράς των επιβατών, κάτι το οποίο έχει επέλθει. Δεν πρέπει να περιμένουμε να ανοίξει η αγορά και γι' αυτό νομίζω ότι οι διατάξεις της αναδιατύπωσης θα βοηθήσουν για το άνοιγμα των αγορών. Προτείνω λοιπόν μία σειρά κανόνων έτσι ώστε στο άρθρο 7 να δούμε πώς έχει αυτός ο σύνδεσμος των οικονομικών φορέων και των ρυθμιστικών αρχών. Υπάρχει και μία μεταβατική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας έχω εντάξει αρκετούς κανόνες έχουν ενταχθεί αρκετούς ε, κανόνες για να υπάρχουν εγγυήσεις ως προς την κινητικότητα και το προσωπικό καθώς και τις κοινωνικές ε, ε, ρήτρε και την ασφάλεια και την υγεία στον τομέα. Επίσης, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τις απόλυτα αναγκαίες υπηρεσίες, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η συντήρηση των σειρμών και των σταθμών. Γι' αυτό πιστεύω ότι έτσι και μόνον έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε να μπουν στον τομέα άλλοι οικονομικοί φορείς. Θεωρώ ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να προσελκύσουν πελατεία. Γι' αυτό στο άρθρο 13 υπάρχουν τροπολογίες υπέρ της πρότασης της Κομισιόν, έτσι ώστε να καταστεί πιο σαφές το όλο και να είναι πιο σαφής και η αρχική πρόταση της Κομισιόν. Αυτά είναι τα βασικά σημεία. Βεβαίω είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διασάφηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κυρία Σαρακίνη, θα σας πω πώς έχει ο κατάλογος ομιλητών. Uh,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

Δηλαδή μιλήστε τώρα, διαφορετικά θα παρέλθει ο χρόνος. Δεν μπορεί να γίνει εκ των υστέρων. Τώρα θα επιμερίσω το χρόνο. Πέντε λεπτά για τους σκιώδεις και τρία λεπτά οι υπόλοιποι. Εντάξει. Πέντε λεπτά. Ο κύριος Κούν καταρχήν. E. Ευχαριστώ. Ο χρόνος τρέχει. Ευχαριστώ και την κυρία Σερακιάνη, η που κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες, παρακολούθησε με ανοιχτό πνεύμα την διαδικασία διαβουλεύσεων και ήταν και διατεθειμένη να μας διαθέσει τις απαραίτητες πληροφορίες, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για το δύσκολο αυτό το θέμα. Θέσαμε το ερώτημα όταν η πρώτη δέσμη μέτρων για το σιδηρόδρομο τέθηκε σε ισχύ, γιατί άραγε είχε τόσο λίγη επιτυχία. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Γιατί άραγε οι χώρες μέλη γιατί αντιστάθηκαν τόσο πολύ στο να προωθήσουν περισσότερα εμπορεύματα και επιβάτες με το σιδηρόδρομο και διαμεθοριακά μάλιστα. Και αν εξάσει κανείς τις συζητήσεις του Συμβουλίου είναι πραγματικά χάος. Είναι δύσκολο Ωστόσο, το Κοινοβούλιο μπορεί να επιτύχει σημαντική πλειοψηφία και πρέπει. Για παράδειγμα, η διάρθρωση της χρηματοδότησης, επενδύσεις στο σιδηρόδρομο, διαλειτουργικότητα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη ώστε να πέσουν οι φραγμοί αυτοί. Είδαμε και ξαναείδαμε συζητήσεις πάνελ το τελευταίο καιρό και διαρωτηθήκαμε πού είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες της ε, φιλελευθεροποίησης στο unbundling δεν μιλώ για το κόστος σήμερα αλλά και στο μοντέλο holding γι' αυτό δεν θα πρέπει να μείνουμε μοναχά στο μοντέλο της υποδομής για να δούμε αν θα επιτύχει η απελευθέρωση Αυτά νομίζω τα έχουν δείξει και οι συζητήσεις και μέσα στις πολιτικές ομάδες αλλά και μέσα στις χώρες μέλη που δίνουν μια κατεύθυνση και που δείχνουν ότι σωστό θα ήταν να υπάρξει και ανταγωνισμός ανάμεσα στα δύο μοντέλα αλλά υπό τις ορθές συνθήκες και εκεί η διαφάνεια είναι το α και το ω. Πρέπει να είναι σαφέστατα, ε, σαφέστατο μάλλον η κυριότητα τι σημαίνει. Οι τροχιές, οι σηματοδότες, η, τα κτίρια των σταθμών και ο υπολογισμός πρέπει να είναι σαφής, ώστε κάθε ανταγωνιζόμενος μέσα στην Ευρώπη να μπορεί να ανταγωνιστεί με ξεκάθαρους όρους ανταγωνισμούς. Και ποιος μπορεί να εξασφαλίσει αυτή την διαφάνεια, όχι βεβαίως, όχι βεβαίως κάποιος ο οποίος βρίσκεται μέσα σε μια holding εταιρεία, αλλά μόνο το ρυθμιστικό όργανο, η ρυθμιστική αρχή. Άρα πρέπει να είναι ένα όργανο το οποίο να διαθέτει και προσωπικό και εξοπλισμό και αρμοδιότητες και να μπορεί να πει «Ιδού, λαμβάνω μια αίτηση, γίνεται δεκτή γιατί είναι σύμφωνη με, τους, με τις ρυθμίσεις ή απορρίπτεται διότι και ούτω καθεξής». Πρέπει να υπάρχει σαφήνεια λοιπόν, διαφάνεια μάλλον. Η απορριπτεται διοτι και ουτω καθεξης πρεπει να υπαρχει αφηνεια λοιπον διαφανεια μαλλον η λειτουργια του δικτύου που συνήθως είναι κρατική επένδυση και ανάμεσα στις μεγάλες ε, επιχειρήσεις και μεγάλους ομίλους τι ροές κονδυλίων υπάρχουν τότε θα υπάρξει απόλυτη σαφήνεια και θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Ένα άλλο κύριο σημείο είναι οι υπηρεσίες. ο καθένας μπορεί να είναι υπέρ του unbundling, του διαχωρισμού δηλαδή της εκκλησίας από την χρήση, κατά, ιδιωτικοποίηση όχι και βεβαίως να βγει και να τα πει. Αλλά δεν είναι αυτό το κρίσιμο σημείο. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς θα ανοίξουμε την αγορά. Και εδώ εντάσσονται και οι υπηρεσίες. Είτε θα συνδεθεί τώρα με κάποιο δυναμικό, δηλαδή θα πούμε 20% πρέπει να μένει ανοιχτό και use it or lose it, χρησιμοποίησε το μη κινδυνεύει το χάσεις και φοβάμαι ότι θα χάσω και, χρόνο, και το χρόνο αγόρευσής μου τώρα σιγά σιγά για τη διαλειτουργικότητα είπαμε νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε ένα καλό μοντέλο και θα μπορέσουμε να προωθήσουμε και καλές συμβιβαστικές λύσεις με συνύπαρξη των δύο συστημάτων ώστε να υπάρξει περισσότερη απελευθέρωση, περισσότερος ανταγωνισμός ώστε επιβάτες να μπορούν να πάνε από τη Βαρσοβία μέχρι το Παρίσι ή το Λονδίνο και από τις σκανδιναβικές χώρες μέχρι τη Ρώμη χωρίς προσκόμματα. Και το ίδιο να ισχύει βέβαια και για τα εμπορεύματα. Ευχαριστώ κύριε Κούν. Ο κύριος Τρεμόλσκι. Ευχαριστώ ε, πρώτα την εισηγήτρια για την δουλειά που έκανε καθώς και την ομάδα της, δηλαδή το προσωπικό της, καθώς και τους δικούς μου που με συνέδραμαν σημαντικά. Πρώτα πρώτα για το unbundling. Η ομάδα των φιλελευθέρων δεν είναι υπέρ της πλήρους αποσύνθεσης του πλήρους unbundling. Όπως είπα και στις συζητήσει μας, δεν υπάρχει σαφή συσχετισμό μεταξύ ανταγωνισμού, ανταγωνισμού και των διαρθωτικών δομών. Εάν επιβάλλουμε τώρα την υποχρέωση διαχώρησης, αποσύνδεσης δεν θα έχουμε δυσανάλογο κόστος με την αποτελεσματικότητα. Ας αναμείνουμε λοιπόν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Μπορούμε να περιλάβουμε μια τελογική σκέψη με την παραπομπή ότι αναμένουμε την έκδοση της νομολογίας του δικαστηρίου για το θέμα αυτό. Ωστόσο, είμαστε ανοιχτοί για να δούμε πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ανεξαρτησία του διαχειριστού της υποδομής. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να, να μπορούσαμε να πούμε ότι τα μέλη του Δυτικού Συμβουλίου της Holding δεν, κάθονται, δεν βρίσκονται και δεν είναι και μέλη του Δυτικού Συμβουλίου της ε, ε, εταιρεία που διαχειρίζεται την υποδομή. Μπορούμε να ανοίξουμε την εσωτερική αγορά για τους επιβάτες εκτός του PSO. Και σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στις αγορές, τροπολογία 9, θεωρούμε ότι το Regulatory Department της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να υποστηρίξει τους αρμόδιους εθνικούς οργανισμούς ώστε να ενισχύσουν την πρόσβαση στην αγορά της, ε, του σιδηροδρόμου. Σε αρμόδιες γενικές διευθύνσεις, MOVE και Competition της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορούν να συμμετάσχουν μέλη τους σε ένα ειδικό όργανο το οποίο θα ε, κάνει αυτή τη δουλειά. Και εδώ τροπολογία 80 τη εισηγήτρια. Αυτό το Regulatory Department τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρεμβαίνει μόνο εάν η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή δεν το πράττει σε περίπτωση ε, διαφορών. Όσο πιο ισχυρός, όσο πιο ισχυρός θα είναι ο οργανισμός αυτός, τόσο πιο ανοιχτή θα είναι η αγορά. Γιατί βεβαίως όλοι οι εθνικοί οργανισμοί ρύθμισης δεν είναι ισοδύναμοι σε ό,τι αφορά ε, προσωπικό και δυναμικό κλπ. Και γι' αυτό περιλαμβάνω εγώ και μια τροπολογία που θα λέει ότι θα πρέπει να συνδέονται αυτά απολύτω με τι ανάγκε τη αγορά. Ταυτόχρονα μπορούμε να ενισχύσουμε την τροπολογία 11 προσθέτοντας ότι ο Ευρωπαϊκό Regulatory Body θα πρέπει να, με αυτού να προηγηθεί το Regulatory Department της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίσης στα άθρα 56 και 57 οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές που δεν ασέβονται προθεσμίες και εντολή τους θα πρέπει να παραπέμπονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά την ελάχιστη ασφάλεια, μάλλον την ασφάλεια των ελάχιστων εισφορών, θέλουμε επίσης να ζητήσουμε από τις εθνικές, από τα εθνικά κοινοβούλια να ζητήσουν ενίσχυση των οργάνων αυτών. Και σε ό,τι αφορά την τροπολογία 88, εμείς θα θέλαμε να είμαστε περισσότερο φιλόδοξοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή θα πρέπει μέχρι το τέλος του 2012 να καταθέσει πρόταση για το Ευρωπαϊκό Regulatory Body. Επίσης, του χρόνου προβλέπεται αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να υποβάλει πρόταση για το άνοιγμα των εσωτερικών αγορών μεταφοράς επιβατών. Να περιληφθεί λοιπόν και αυτό στην συζήτησή μας. Σε ό,τι αφορά τις ελάχιστες προσφερόμενες υπηρεσίες σε περίπτωση απεργίας, εμείς δεν θέλουμε να διαγραφεί αυτή η δυνατότητα. Απεργία σε μια χώρα δεν θα πρέπει να μπλοκάρει την κίνηση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό των, α, του άμεσου κόστους, τροπολογίες 118 έως 120, να βάλουμε και συντάξεις και kindergarten ως άμεσο κόστος. Αυτό όμως θα κάνει τα τρένα πιο ακριβά, αν δεν είναι ανταγωνιστικά. Και για την τροπολογία 121 δεν είμαστε υπέρ να ε, διαγραφεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναγνωρίζουμε ότι δεν έχουν το ίδιο ενδιαφέρον όλες, ε, όλα τα μερίδια της, όλοι οι της αγοράς για όλες τις χώρες μέλη. Και ο ρυθμιστικός οργανισμός θα μπορεί να παρεμβαίνει εκ των υστέρων μόνο σε περιπτώσεις διαφορών και καταγγελιών. Τέλος, άρθρο 66, σε ό,τι αφορά την μεταφορά της αναδιατύπωσης στο εθνικό δίκαιο. Το Συμβούλιο θα ζητήσει διετία για την εφαρμογή της οδηγίας. Ορισμένες χώρες μέλη ζητούν 3 έως 5 χρόνια. Αυτό δεν είναι αποδεκτό. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να επιμείνει στον ένα χρόνο, στο ένα έτος. Ευχαριστώ. Κράμερ, 5 λεπτά από τους πράσινους. Ευχαριστώ και εγώ για την έκθεση που έχει γίνει βέβαια πλέον τώρα η συζήτηση πιο συγκεκριμένη από τις, τις προηγούμενες συζητήσεις. Κάτι με απογοητεύει. Όλοι βέβαια θέλουμε ενιαίο σιδηροδρομικό δίκτυο σε όλη την Ευρώπη και ανταγωνισμό χωρίς διακρίσεις. Συμφωνούμε. Εάν εξετάσουμε τότε το ευρωπαϊκό τοπίο, η βασική διαφορά έγκυται όχι στο αν είναι χωριστή ή όχι, αποσυνδεδεμένη ή όχι η οχι αποσυνδεμενη η γιατί υπάρχουν χώρε που έχουν κάνει την αποσύνδεση αλλά είναι closed shop και είναι άλλε που δεν το έχουν κάνει και είναι ανοιχτέ. Εμεί θέλουμε ανοιχτό δίκτυο για όλου, αλλά υπό έντιμου όρου ανταγωνισμού. Και γι' αυτό δεν αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο επιμένετε στην έκθεσή σα. τόσο πολύ για αυτό το περίφημο unbundling, ενώ γνωρίζουμε ότι δεν είναι αυτό το αποφασιστικό κριτήριο. Μπορούμε να επιβάλλουμε το unbundling σε όλες τις χώρες, παρόλα αυτά οι συνθήκε δεν πρόκειται να αλλάξουν, διότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν άλλοι παράγοντε οι οποίοι είναι κρίσιμοι. Εγώ ω πράσινο είμαι υπέρ τη αποσύνδεση τη ιδιοκτησίας από την διαχείριση του δικτύου, αλλά δεν είναι το απαραίτητο κριτήριο. Και είχαμε συμφωνήσει επίση ότι ο ρυθμιστικό οργανισμό είναι κρίσιμου ρόλου οι χώρες οι οποίες έχουν ανεξάρτητο regulatory body έχουν και το άνοιγμα των δικτύων και επομένως οι αποφάσεις λαμβάνονται ταχύτερα. Γι' αυτό και δεν κατανοώ για ποιο λόγο παίρνετε την απόφαση της Κομισιόν ότι δηλαδή μέσα σε τέσσερις εβδομάδες σε κάθε περίπτωση, in any case, θα πρέπει να, να αποφασίζετε αν θα έχω το λεγόμενο slot. Λέμε πάλι καταρχήν, λέτε πάλι καταρχήν εκεί, στη χώρα σας μέσα σε δύο μήνες λαμβάνεται απόφαση εάν κανείς θα έχει σλότ ή όχι, χρονοθυρί δηλαδή ή όχι. Εφόσον όμως έχει σωστά συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο. Αν κάποιος έχει κάνει λάθος το ερωτηματολόγιο φτάνει να περάσουν και δύο χρόνια και δεν λαμβάνει απάντηση. Υπάρχουν άλλες χώρες που έχουν regulatory body και δεν λαμβάνουν απάντηση ακόμα και αν περάσουν τα δύο χρόνια και είτε έχουν συμπληρώσει είτε όχι το ερωτηματολόγιο. Εγώ λέω, εν πάση περιπτώσει πρέπει να λαμβάνετε απάντηση μέσα σε τέσσερις εβδομάδες και μετά μπορούμε να το συζητήσουμε εάν η απόρριψη, η απόρριψη είναι ένομη ή όχι. Γιατί βεβαίω μιλάμε μόνο για την απόρριψη της αίτηση. Μια νέα ή μια μικρή επιχείρηση η οποία ακόμα μετά από μια διετία δεν γνωρίζει εάν θα έχει πρόσβαση στο δίκτυο, δεν πρόκειται βεβαίω να αγοράσει μηχανέ έλξη, ούτε οχήματα, ούτε να κάνει καμιά άλλη επένδυση. Γι' αυτό ο το ρυθμιστικό όργανο είναι το κρίσιμο σκαλί και πρέπει αυτό να αποφασιστεί να εγκριθεί. Εσεί κύριε Κούν επίση είπατε ότι η διαφάνεια είναι απόλυτα απαραίτητη. Από πού προέρχονται τα κονδύλια και πού πηγαίνουν. Θέλουμε βέβαια τα κονδύλια που πάνε για υποδομές να πάνε εκεί όπου που ήρθαν. Και θέλουμε για υποδομέ να πανε εκει οπου που ηρθαν και έντιμους και έντιμου όρου ανταγωνισμου Δεν είναι δυνατόν, το είπα και την προηγούμενη φορά, στην Γερμανία, στο Βερολίνο, να είναι διπλάσιο το κόστο ε, για την χρήση ενό τμήματο του δικτύου από την είναι και στο Αμβούργο πάλι είναι διπλάσιο από την ε, Βόρεια Ρινανία. Πρέπει να είναι εξασφαλισμένο ότι θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν τα δίκτυα, διότι οι χώρες μέλη τα έχουν χτίσει τις υποδομές αυτές επί δεκαετίες και τις έχουν διαχειριστεί και τώρα πρέπει να τις ανοίξουν στον ανταγωνισμό. Ε, τώρα, για τον θόρυβο και για το EATMS έχετε διαφορετικές τιμές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 5% μείωση δεν είναι βέβαια κανένα ιδιαίτερο κίνητρο για να μειωθεί ο θόρυβος των ε, σειρμών. Αλλά για το EATMS το σύστημα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της πραγματικότητας. Είναι ρεαλιστικό. Διότι ανταγωνίζεται και με τις συχνότητες που χρησιμοποιούμε και για άλλα πράγματα, για παράδειγμα τα για τα κινητά τηλέφωνα. Όταν μαθαίνω τώρα ότι όλες οι σιδηροδρομικές εταιρείε στην Ευρώπη τονίζουν την σύγκρουση αυτή και έρχεται ωστόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει ότι για τρία χρόνια δεν θα κάνουμε απολύτω τίποτα, τότε δεν αντιλαμβάνεται η Κομισιόν ποια είναι η ανάγκη. Υπάρχουν ακόμα βέβαια πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν, ούτε και μπορώ να μιλήσω τόσο πολύ, αλλά για την ασφάλεια, για την ασφάλιση δηλαδή. Γιατί το ανώτατο όριο είναι 100 εκατομμύρια, ενώ μπορεί να υπάρξει διαφορά και μεγαλύτερη. Γιατί βάζετε ανώτατο όριο. Εγώ ξέρω ότι οι ασφάλειες βάζουν ένα κατώτατο όριο. Και για το ανώτατο όριο εξαρτάται από τι είδους ασφαλιστική σύμβαση κάνετε. Διότι εν τέλει με αυτά που λέω μόνο έτσι θα έχουμε ένα κοινό δίκτυο σιδηροδρομικό όπου καθένας θα μπορεί να μετακινείται με αυτό και αυτό είναι προς το συμφέρον των επιβατών, των πελατών. Αυτό θέλουμε να επιβάλλουμε στην Ευρώπη και γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα αυστηρό ρυθμιστικό οργανισμό. Ευχαριστώ κύριο Ζήλε. Πέντε λεπτά. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πολύ δύσκολη εργασία στην οποία χρειάστηκε να αντεπεξέλθει. Ήταν πολύ δύσκολη η εργασία που είχε επιτελέσει. Πολλά από τα βασικά σημεία έχουν καλυφθεί, αλλά στην τροπολογία 55 στο θέμα της ασφάλισης μιλάτε για μέγιστη και ελάχιστη κάλυψη και μιλάτε για μέγιστη κάλυψη 100 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος. Αυτό όμως δεν καλύπτει όλες τις καταστάσεις γιατί έχει μεγάλη σημασία η εμβέλεια του ατυχήματος. και βεβαίως ανάλογα και με την ταχύτητα η, πολιτική της, η ασφαλιστική πολιτική είναι διαφορετική. Υπάρχουν τέσσερις χώρες που έχουν ένα διαφορετικό πλαίσιο. Μεταξύ αυτών εντάσσεται και η Φιλανδία γιατί εμείς συνδεόμαστε με το ρωσικό σιδηροδρομικό δίκτυο θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη και αυτή την πτυχή. Και ως προς την ε, καταβολή της αποζημίωσης θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το πλαίσιο. Θα πρέπει να απλουστεύσουμε αυτό το σύστημα έτσι ώστε κάθε τμήμα, κάθε segment να αποφασίσει ποιοι κανόνες θα ισχύουν. Δηλαδή να υπάρχουν ελάχιστα και μέγιστα όρια. Ως προς τη ρυθμιστική αρχή υποστηρίζω την ε, ιδέα ότι μια ρυθμιστική, η ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να είναι πιο ισχυρή σε κάθε κράτος μέλος, αλλά και ο Ευρωπαίος ρυθμιστής θα πρέπει να έχει συγκεκριμένα καθήκοντα. Αν δείτε την τεχνολογία των πληροφοριών στα 27 κράτη-μέλη, βλέπετε ότι ίσως αυτή θα ήταν η καλύτερη κατεύθυνση που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Δεν ε, νομίζω ότι χρειάζεται ένα νέο ρυθμιστικό όργανο σε αυτή τη φάση των εργασιών. Αλλά θα πρέπει ο εκπρόσωπος, ο ρυθμιστής, να μπορεί να παρευρίσκεται σε συναντήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως, οι ρυθμιστικοί οργανισμοί, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να ασχολούνται με τα διάφορα, με τα επιμέρους segments, με τα επιμέρους τμήματα. Όταν μιλάμε για παρόχους υπηρεσιών, το θέμα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και θα ήθελα η συγκήτρια να προβάλλει ένα συμβασμό, διότι όπως είπε και κάποιος άλλος συνάδελφος, υπάρχει διχογνωμία και θα πρέπει να βρούμε ένα μέσο όρο. Ευχαριστούμε κυρία Βίλς για πέντε λεπτά. Frau ähm, der von Ihnen vorgelegte Entwurf eines Berichts teilt in seiner Begründung. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ότι η προσέγγιση της κυρίας ε, Σαρακιάνη ε, είναι πολύ κοντά σε αυτή την... Ε, της Κομισιόν. Αλλά πέρσι είχαμε την εντύπωση ότι δεν υπήρχε επαρκής απορρίθμιση ή ιδιωτικοποίηση στον τομέα των συνδυροδρόμων Και σε μία ακρόασή μας στις, 13, στις 3 Μαρτίου με εμπειρογνώμονες από το τομέα των σιδηροδρόμων κατέδειξε ότι το στάδιο απελευθέρωσης και ιδιωτικοποίησης οδήγησε σε χαμηλότερες ποιοτικές προδιαγραφές είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση χάους του διαδρόμους. Επίσης είχαμε πολλά ατυχήματα στην Ιταλία, στη Σαξονία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και ως προς τις... την αιτιολογική σκέψη δεν γίνεται μνήα σε ένα βασικό σημείο, το δικαίωμα απεργίας και πιστεύω ότι εάν παραβιάζουμε αυτό το δικαίωμα, αυτό ε, προσβάλλει όχι μόνο το τομέα των σιδηροδρόμων, αλλά όλους τους ε, τομείς. Η τροπολογία 117 είναι μια τροπολογία την οποία θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε. Χρειάζονται ελάχιστα επίπεδα λειτουργίας όταν μιλάμε για δικαίωμα απεργίας. Αυτό όμως θα έπρεπε να απομακρυνθεί από την οδηγία. Ως προς τους παρόχους υπηρεσιών, συμφωνείτε με την Επιτροπή, αλλά νομίζω ότι σφάλετε. Διότι είδαμε ότι πολλές ε, επιχειρήσεις οδηγήθηκαν στην εξωτερική ανάθεση εξυπηρέτηση, στο outsourcing και αυτό μειώνει και τα δικαιώματα των εργαζομένων σε αυτό τον τομέα. Συρρυκνώνει τα δικαιώματα των ε, εργαζομένων ως προς τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξης από την αιτιολογική σκέψη και μόνο δεν καταλαβαίνω ποια είναι η θέση της εισηγήτριας. Θα ήθελα να πω από τη δική μας άποψη ότι απορρίπτουμε τις κατεξιοδότηση πράξεις ε, όπως ορίζονται. Ίσως θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη τα παραρτήματα περισσότερο, γιατί νομίζω ότι δεν επιτρέπουν ε, οι πράξεις αυτές να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι από νομικής και δημοκρατικής άποψης υπάρχει θέμα δημοκρατικού ελέγχου και εποπτείας θα πρέπει να γίνει μια συνολική αξιολόγηση. Οι ρυθμιστές δυστυχώς περιορίζουν την εμβέλεια λειτουργίας και θα σταθώ εδώ γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε. Επόμενος, για τρία λεπτά, ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμείς στηρίζουμε όσον αφορά την αρχή, την ελευθέρωση των σιδηροδρόμων. Θέλω όμως να επιστήσω την προσοχή σας σε κάποιες ιδιαιτερότητες που ισχύουν για τη Λιθουανία και που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη. Εμείς έχουμε μεγαλύτερο δίκτυο από τις άλλες χώρες και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ενταχθούν οι δικοί μας σιδηρόδρομοι στους ε, σιδηρόδρομους, στο σύστημα σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 75% όλων των σιδηροδρομικών μεταφορών γίνεται ε, από εμπορικούς σιδηροδρόμους από τρίτες χώρες. Και δεν θα ήταν καθόλου σοφό να εφαρμόσουμε τα τέλη αυτά σε ε, πάρχους από τρίτες χώρες που δεν καλύπτει, το κόστος δηλαδή που δεν καλύπτεται στο εσωτερικό της χώρας από τους ε, ντόπιου. Δεν είναι σωστό να καλύπτεται μόνο το 35% του κόστους όπως προτείνεται. Γιατί αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνησή μας θα έπρεπε να καλύψει το υπόλοιπο κόστος. Ε, τα τέλη υποδομών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ολόκληρο το κόστος των φορέων και οι τρίτες χώρες δεν επιδοτούν τις εμπορικές μεταφορές μέσα από τη Λιθουανία, που περνάει μέσα από τη Λιθουανία δηλαδή. Γι' αυτό και προτείνουμε στο άρθρο 31, στο σημείο 3 ή στο 32, στο σημείο 1, να υπάρξει κάποια ένδειξη που να λέει ότι τα τέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόλοιπα υπόψη την κατάσταση των χωρών ε, αυτών που έχουν μεγαλύτερο μέρος τέτοιου εμπορίου. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γκρός, τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσεγγίσω τη σημερινή συζήτηση με πιο σφαιρικό τρόπο. Στο Λαϊκό Κόμμα έχουμε καταθέσει και έχουμε συζητήσει βέβαια και με το σκιώδη συγητή μας τις σχετικές τροπολογίες αλλά και η σημερινή συζήτηση έχει ενδιαφέρον, διότι νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας δύο θέματα όπου το Συμβούλιο στο παρελθόν είχε δείξει συμφωνία, όπου τώρα όμως δεν είναι πλέον, δεν δείχνει καμία διάθεση να εφαρμόσει τα όσα ήδη έχουν εγκριθεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό και τίθεται τώρα καταρχήν το ερώτημα σε όλα τα έγγραφα των τελευταίων εβδομάδων και μηνών και ετών διαπιστώνουμε ότι ο σιδηρόδρομος καλείται να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί όμως οι οποίοι καλούνται να δώσουν τα κονδύλια δεν επιθυμούν να βελτιώσουν τις υποδομές, δεν επιθυμούν να τις επεκτείνουν, καθώς επίσης και οι αρμόδιοι νομοθέτες δεν θέλουν να εγκρίνουν σχετική νομοθεσία. με αυτήν την συζήτηση πρέπει να συνδεθεί και μια συζήτηση γύρω από τις υπηρεσίες και την προσφορά υπηρεσιών. Πράγματι ο σιδηρόδρομος σε πολλές χώρες προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες είναι εκτός ανταγωνισμού και θα πρέπει να παραμείνουν και στο μέλλον εκτός ανταγωνισμού που σημαίνουν όμως απασχόληση και όπου το καθεστώς των απασχολουμένων εμπλέκεται στην σύγκρουση αυτή την οποία αντιμετωπίζουμε μπροστά μας. Γι' αυτό τα θέματα αυτά πρέπει να τεθούν ανοιχτά και όχι να γίνεται προσπάθεια να, να προστατευτεί η απασχόληση και το καθεστώ της απασχόλησης αυτής με άλλα μέσα τα οποία αποβαίνουν εν τέλει σε βάρος της αγοράς. Εδώ διατίθεται σημαντικά δημόσια κονδύλια και για την, και για την προσφορά υπηρεσιών αλλά και για τις υποδομές και μάλιστα και για παρόχους υπηρεσιών που δεν βρίσκονται μέσα στα πλαίσια των σιδηροδρόμων. Γνωρίζουμε δηλαδή παρόχου υπηρεσιών οι οποίοι προσφέρουν όχι μόνο μεταφορά σιδηροδρομική αλλά και αλλού. Άρα η διαφάνεια των χρηματικών ροών είναι απόλυτα απαραίτητη διότι δεν είναι δυνατόν αύριο δημόσια κονδύλια να χρησιμοποιούνται έμεσα για να υποσκάπτεται ο ανταγωνισμός. Γι' αυτό και είμαι απόλυτα σύμφωνος με το ότι ο ρυθμιστής αύριο θα κληθεί να παίξει τον σημαντικότερο ρόλο. Και αν δεν δώσουμε όλα τα μέσα, όλα τα όπλα στον ρυθμιστή, όχι ρυθμίζοντας και την τελευταία λεπτομέρεια, αλλά αν δεν του δώσουμε όλα τα μέσα στον ρυθμιστή για να παίξει τον ρόλο του, δηλαδή να κάνει τον έλεγχο της διεξαγωγής Ο ρυθμιστής θα εξετάζει εάν οι τιμές είναι σωστές, εάν οι προσβάσεις είναι σωστές, αν δεν υπάρχουν δηλαδή τεχνικά ή άλλα κολλήματα. Αυτά είναι τα σημαντικά κατά τη γνώμη μου. Και ο ρυθμιστής αυτός, εφόσον εμείς εννοούμε τα πράγματα αυτά σοβαρά και θέλουμε πράγματι αύριο να έχουμε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο, δεν θα κληθεί μονάχα να φτιάξει ευρωπαϊκό δίκτυο αύριο, αλλά θα χρειαστεί ε, να γίνει από σήμερα. Έχουμε ήδη δίκτυα τα οποία λειτουργούν διαμεθοριακά. Γιατί λοιπόν όχι και στον τομέα αυτό. Εάν γίνει δεκτό ότι ο ρυθμιστής αύριο θα μπορεί να, δραστηριοποιηθεί, να δραστηριοποιείται και στο, στο ε, ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βεβαίως θα κάνουμε και άλλες προτάσεις. Ευχαριστώ κύριε Γκρός. Ελ Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ την εισηγήτρια. Όντω με επιστημονικό τρόπο εξετάζει το θέμα τη, Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς όμως πιο πολύ είναι πώς θα έχουμε ανταγωνιστικούς σιδηροδρόμου και πώς θα τραβήξουν περισσότερα ε, πορεύματα από τις οδικές μεταφορές και πώς θα είναι πιο αποτελεσματικοί. Το θέμα της ε, συμβατότητας, της τεχνικής συμβατότητας είναι κάτι που μας απασχολεί όλος ιδιαίτερος και βέβαια και η χρηματοδότηση των υποδομών και των υπηρεσιών. Αυτό το θέμα είναι ένα θέμα που συνδέεται άμεσα με την αγορά και επικεντρώνεται στο θέμα της νομοθετικής ρύθμισης. Νομίζω ότι είναι μια καλή απόφαση να επικεντρωθούμε σε αυτό και να μην μπούμε σήμερα στη συζήτηση για την ελευθέρωση των εθνικών μεταφορών. Έχουμε χρόνο γι' αυτό στο μέλλον αυτό που είναι βασικό είναι ο ρυθμιστής να έχει χρόνο να μπορέσει να παρέμβει και να μπορέσουμε έτσι να στηρίξουμε τις προτάσεις της εισηγήτριας. Υπάρχει ένα δίκτυο, πάντως συμφωνώ με τον κύριο Γκρός, ο οποίος λέει ότι ίσως πρέπει να πάμε λίγο ακόμα πιο μακριά και να δούμε μήπως το έμβριο να μπορέσουμε να το προχωρήσουμε και να έχουμε μια ευρωπαϊκή ρύθμιση με τους λεγόμενους διαδρόμους μεταφορών, τους corridors. Αυτό πρέπει να ερευνηθεί περισσότερο. Πάντως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι εμείς δεν έχουμε καταλήξει οριστικά ως ομάδα. Σημειώνουμε την πρόταση της εισηγήτριας πρέπει να συζητήσουμε μεταξύ μας, να εξετάσουμε σε βάθο τις προτάσεις αυτές. Αυτό πάντως που μένα με ενδιαφέρει είναι το σύστημα αυτό να είναι λειτουργικό, να λειτουργήσει, να έχουμε έτσι μια καλή τίμια αγορά με θεμητό ανταγωνισμό που θα ε, βοηθήσει να έχει κάποιο μέλλον ο τομέας των σιδηροδρόμων και να είναι ανταγωνιστικός. Αυτό μας ενδιαφέρει γιατί η σημερινή πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει καλός ανταγωνισμός Το θέμα είναι το κατά πόσο πρέπει να δούμε τις υποδομές ανεξάρτητα, να λειτουργούν ανεξάρτητα από την ε, λειτουργία των σιδηροδρόμων. Σίγουρα χρειάζεται διαφάνεια και κάτι παραπάνω. Πρέπει να προσπαθήσουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, ληφθεί υπόψη δικιά μας η θέση. Έχω εδώ πέρα και διάφορες άλλες λεπτομέρειες Πρώτον το θέμα του κοινωνικού παράγοντα. Είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας τους εργαζόμενους, ό,τι κάνουμε δηλαδή να μην αποβεί σε βάρος τους. Η εισηγήτρια πρέπει να συμπεριλάβει αυτό το σημείο του κοινωνικού παράγοντα για τους εργαζόμενους. Επίσης το τελευταίο που θέλω να θίξω εδώ είναι το θέμα της χρηματοδότησης. Συμφωνώ ότι πρέπει από τα κράτη-μέλη να έρθουν τα χρήματα για να στηριχτεί ο τομέας. Γι' αυτό και πρέπει να δούμε το θέμα του άμεσου κόστους για την υποδομή, πώς θα οριστεί, να οριστεί καλά και να κάνουμε και μία ανάλυση για το τι μπορούμε να πετύχουμε στα διάφορα κράτη-μέλη όσον αφορά τις υποδομές. Αυτά. Αργότερα θα επανέλθουμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μάση έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ με τη σειρά μου την κυρία Σερακιάνη για την σε βάθος και θαραλέα εργασία της διότι βεβαίως λαμβάνει άλλη θέση από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με αυτόν τον τρόπο έρχεστε βέβαια να ρίξετε και περισσότερο βάρος στο λεγόμενο unbundling το οποίο βέβαια ενδεχομένως θα είχε και ε, να αντιμετωπίσει και διαφορές απόψεων και εδώ στο Κοινοβούλιο. Πάντως το βρίσκω θαραλέο αυτό. Βέβαια, όπως έχετε τροποποιήσει το κείμενό σας, νομίζω δεν βρίσκεται πλέον στον σωστό δρόμο που χρειαζόμαστε για να έχουμε περισσότερο ανταγωνισμό, αλλά και περισσότερη πρόσβαση. Διότι αυτό είναι ο στόχο. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε την ευρωπαϊκή αγορά. Χρειαζόμαστε βεβαίω περισσότερη διαλειτουργικότητα και αυτό σωστό είναι. Χρειαζόμαστε όμω και να υπάρχει πρόσβαση παντού για όλου του φορεί οι οποίοι θέλουν να μεταφέρουν κάτι τι μέσω σιδηροδρόμου. Γι' αυτό και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον αγαπητό φίλο Μιχαήλ Κράμερ Βέβαια δεν συμφωνούμε και πάντα εμείς οι δυο, αλλά έχει δίκιο. Χωρίς αυτό να έχει, ε, χωρίς να έχει ε, απαραίτητα ως λόγο το ότι είμαστε και οι δύο Γερμανοί και εκεί το σύστημα λειτουργεί. Αλλά στην περίπτωση αυτή νομίζω απλώς είμαστε και οι δύο ευφύς άνθρωποι και διερωτώμεθα πώς μπορούμε με τον καλύτερο τρόπο να επιτύχουμε τον τελικό στόχο της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Και εκεί θεωρώ ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κινείται περισσότερο προς την κατεύθυνση αυτή. Βεβαίως, ε, από σύνδεση ιδιοκτησίας από διαχείριση είναι σωστή. Και στη Γερμανία όπου υπάρχει πολλή κίνηση ε, από το σιδηρόδρομο χρειάζεται ωστόσο και εκεί ακόμα βελτίωση. Χρειαζόμαστε λοιπόν να ρυθμιστεί ο οποίο θα είναι ισχυρός. Χρειάζεται να συζητήσουμε και για τέλη που είναι άλλη υπόθεση από την ε, υπόθεση αυτή και όπως είπε ο κ. Στεμόλη και εξ, ονόματο τη της ομάδας μου προς αυτή την κατεύθυνση να κινηθούμε. Ευχαριστώ. Ρικέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια και από μένα και δεν το λέω έτσι τυπικά. Θέλω πραγματικά να συγχαρώ την κυρία Σαρακιάνη για μια εξαίρετη και πολύ θαραλέα έκθεση και πολύ γερή. Από το θέμα ήταν περίπλοκο. Δεν θέλω να αναφερθώ στα διάφορα μέτρα ένα προς ένα. Δεν νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε τώρα. Αλλά να αναφέρω μερικά γενικά στοιχεία. Δεδομένου ότι πολλές χώρες μέλη πάνε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και παραβιάζουν τις συνθήκες αντί να εφαρμόζουν ήδη την πρώτη οδηγία, δυστυχώς καταλαβαίνω ότι είναι μάλλον αποφασισμένοι να διάσουν από κάθε περιεχόμενο την μέχρι τώρα ρύθμιση, δυστυχώς. Αν λοιπόν χάσουμε το ραντεβού αυτό, πόσο θα υποστηρίξουμε τις οικονομίες στην ενέργεια, την μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα κλπ. Και πώς θα ανοίξουμε την αγορά μας. Ποια είναι τα μέσα για να πετύχουμε. Είναι ακριβώς να αποσυνδέσουμε τις υπηρεσίες από τις υποδομές. Καμία χώρα δεν έχει κάνει αυτή την αποσύνδεση μέχρι τώρα. Και γι' αυτό και υπάρχουν τόσες πολλές δυσκολίες. Όλοι χαίρονται πολύ για το δικό τους εθνικό σύστημα και κανείς δεν θέλει να αλλάξει τίποτα. Χρειάζεται όμως επίσης όρις ε, πρόσβαση στις υποδομές. Η διαχείριση να γίνεται με δυνατότητες χρηματοδότησης αντίστοιχες των αναγκών. Χρειάζεται θάρρος και επενδύσεις από τις χώρες μέλη, να βοηθήσει και η Ευρώπη βέβαια, και να βασιζόμαστε σε μια καλή ρύθμιση από την Ευρώπη για τελειώς πώς θα ε, πετύχουμε την διαχείριση ό,τι διαφωνιών ε, προκύψουν σε διεθνές επίπεδο. Κάναμε διάφορες παρατηρήσεις μέχρι τώρα για τις κατεξουσιοδότηση πράξης. Πρέπει να σεβαστούμε επίση και την υποχρέωση για κοινοφελείς υπηρεσίε. και να σεβαστούμε και τους εργαζόμενους και τα δικαιώματα των επιβατών. Ε, όλοι το ξέρουν ότι ακριβώς αυτό θέλουμε να καταφέρουμε, αλλά τα προβλήματα τα έχουμε με τους εθνικούς αντιπροσώπου. Ελπίζω να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τους εθνικούς εγωισμούς. Αλλιώς οι σιδηρόδρομοι για χρόνια θα βρίσκονται στην κόλαση πάλι. Αν θέλουμε να το ξεπεράσουμε αυτό, πρέπει να επιδείξουμε θάρρος. Αλλιώς, αν καθυστερήσουμε, οι σιδηρόδρομοι δεν θα μπορέσουν να κερδίσουν το χαμένο έδαφος. Πρέπει τώρα να αποδείξουμε αν θέλουμε την Ευρώπη με σιδηρόδρομους ή όχι. Σέβομαι και συγχαίρω για το θάρρος της κυρία Σαρακιάνη, αλλά δυστυχώς είμαι εξίσου απεσιόδοξος όπως και αυτή. Ο κύριος τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Τρία σχόλια. Αφού πρώτα συγχαρώ την εισηγήτρια για την δύσκολη δουλειά της. Θα έρθω τώρα σε ένα πρώτο σχόλιο όπου δεν θα συμφωνήσω μαζί της. Ε, το λεγόμενο unbundling που δεν νομίζω ότι είναι και το κυριότερο θέμα που πρέπει να ξεδιαλύνουμε. Υπάρχουν σιδηροδομικά δίκτυα στην Ευρώπη τα οποία λειτουργούν μια χαρά και ωστόσο δεν έχουν υποστεί το λεγόμενο unbundling και το αντίστροφο. Χρειάζεται λοιπόν ένα ορθό καλό σύστημα και νομίζω ότι είναι περισσότερο η ρυθμιστική αρχή εκείνη η οποία θα παίξει ένα φασιστικό ρόλο. Το δεύτερο, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ασφαλώς μπορεί κανείς εντός μιας διετίας ή μάλλον ετία να ε, περιληφθούν και τα εξωτερικά στοιχεία κόστου. Αλλά τότε πρέπει να γίνει αυτό και στι οδικέ μεταφορέ. Θα δούμε αργότερα ότι αυτό δεν γίνεται. Εάν λοιπόν επιβάλλουμε κάτι τέτοιο, τότε πρέπει να δώσουμε έντιμους όρους ανταγωνισμού και στις οδικές και στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Τρίτο σχόλιο. Όταν έρχονται να με, να με δουν ομάδες επισκεπτών, όταν μιλώ στην Αυστρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μου λένε «Μα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο θεματοφύλακας των συνθήκων». Τώρα, με τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε για πρώτη φορά έχουμε πλέον ενιαία ευρωπαϊκή ρύθμιση για το δικαιώμα της απεργίας στη συνθήκη. Πώς είναι δυνατόν να έρθουμε τώρα με απλές ρήτρε σε κάποια οδηγία να το καταργήσουμε. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως αδιανόητο. Και εγώ είμαι απολύτως αντίθετος. Και εάν αυτό ήταν το νόημα της πρότασης αυτής, τότε θεωρώ ότι ορισμένες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν καταδεχθεί από τα λάθος πρόσωπα. Ευχαριστώ κύριε Λάιθφιντ. Στέρξ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο Κουν. Η αγορά. Και τι κάνουμε, τι κάνουμε αν χρειάζεται μια διαχείριση η οποία ανήκει σε κάποια άλλη συνδρομική εταιρεία ή τυχαίνει διαφορετικής διαχείρισης. Πώς το ρυθμίζεις αυτό. Δεν μπορεί ο άλλος να πει όχι, πρώτα εγώ πρέπει να ασχοληθώ με τα δικά μου και μετά». Ή όταν ο ιδιοκτήτης ενό σταθμού λέει «Τα δικά μου τρένα θέλω να βοηθήσω να πουλήσω εισιτήρια για τα δικά μου». Τέτοια πράγματα πρέπει να αποφύγουμε όταν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός. Τα άρθρα 7 και 13 γι' αυτό είναι ζωτική σημασίας για μένα και πρέπει να δούμε τελικά οι βασικές υπηρεσίες πώς θα λαμβάνουν χώρα γιατί αυτές τις έχουμε αφήσει λίγο στην πάντα. η σύνδεση με μια σειροδρομική εταιρεία δεν πρέπει να έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορείτε να εξυπηρετείτε το κοινό. Έπειτα είναι θέμα και πολιτικής προσωπικού και αυτό είναι ένα κομμάτι. Γιατί έχουμε μια ανεξάρτητη πολιτική προσωπικού, τότε από ποιον εξαρτάται, από τη μητρική εταιρεία. Πού μπορεί να οδηγήσει αυτό. Γι' αυτό πρέπει να δούμε περισσότερο τα παραρτήματα 2 και 3. Και τα άρθρα εκείνα που λένε ποιε υπηρεσίε μοιράζονται, πώ και πώς ανεξάρτητε πρέπει να είναι αυτέ. Πιστεύω ότι είναι ζωτική σημασία σε αυτό. Τώρα κάτι άλλο για το οποίο δεν λέμε πολλά είναι το licensing. Σε μια εταιρεία σιδηροδρομική, όχι για το υλικό, και ένας από τους τρόπους με τους οποίους ε, ε, ξεφεύγει μια εταιρεία είναι ακριβώς αυτή η ασάφεια. Η αγορά κλείνει. Πρέπει λοιπόν να λέμε και κάτι για την διεύρυνση της ε, υπηρεσίας αυτής και πώς θα ενισχυθεί για αυτό το σημείο. Γιατί κατά τη γνώμη μου είναι όπως και με την ε, ιατρική. Πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή άδεια. Το ίδιο να κάνουμε και για τους σιδηρόδρομους. Και τέλος, ο ρυθμιστής. Πολύ βασικό. Δεν είναι κακή η πρόταση της Επιτροπής, αλλά και εδώ είναι που δεν συμφωνώ απόλυτα, ίσως δεν έχω καταλάβει καλά. Ο ρυθμιστής δεν πρέπει να κάνει τους λογαριασμούς, πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Να λέει, να, εμείς αυτά έχουμε υπολογίσει και ο ρυθμιστής να βλέπει, ισχύουν, Τέλος, Πρόεδρε. Είμαι υπέρ του unbundling. Το έχω πει και στην κυρία Σαρακιάνη. Δεν θα έχουμε καλούς σιδηρόδρομους στην Ευρώπη αν δεν υπάρχει ανεξαρτησία. Αλλά είναι μια συζήτηση που θα συνεχιστεί δίχως άλλο. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς έχουμε να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα πιο βασικά, αλλά θα έρθει και αυτόν η σειρά του. Ευχαριστούμε κύριε Στέρκ, ο κύριος Σαζάλη, για τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά τη συζήτηση αυτή θα ήθελα να σας επισύρω την ε, προσοχή σε ορισμένα σημεία. Θα πρέπει να δούμε ορισμένα σημεία που έθιξε η ε, Κομισιόν κατά πόσο μπορούν να ληφθούν επαρκώς υπόψη. Γιατί πολλές φορές ε, μπορεί οι σιδηρόδρομοι να μην μπορέσουν να ανταποκριθούν με αυτές τις ε, επιπρόσθετες χρηματοδοτήσεις για ναι. εξοπλισμό εκ των υστέρων. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ζητήσουν άλλους ναύλους από τους επιβάτες. Ως προς το άρθρο 14 θα ήθελα να πω ότι αναφερόμαστε σε νέες διασυνοριακές συμφωνίες. Διαφορετικά θα είναι πολύ υψηλός ο γραφειοκρατικός ε, φόρτος. Νομίζω ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε με τρίτες χώρες διαφορετικά. Θα είναι πολύ δύσκολο αν χρειάζεται προγενέστερη κοινοποίηση προς την ε, Κομισιόν. Θα πρόκειται για μια σχηνοτενή διαδικασία η οποία δυστυχώς θα πλήξει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των σιδηροδρόμων, ιδιαίτερα στις ανατολικές χώρες. Ως προς τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξεις, αυτό μας ενδιαφέρει είναι η εμβέλεια αυτών των ε, πράξεων όπως ορίζονται από την οδηγία, διότι η Κομισιόν έχει το δικαίωμα να τις αλλάξει. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπαλσάιτης για τρία λεπτά. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για αυτή την εξαιρετική εργασία. Εγώ εργάστηκα σε αυτό το τομέα για πολλά χρόνια και θα ήθελα να πω ότι κατανοώ την εισηγήτρια. Εδώ μιλάμε όχι μόνο για χρηματοοικονομικά θέματα, αλλά και για πολιτικά. Ως προς το μελλοντικό σύστημα σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Μίλησα με συναδέλφους από τα βαλτικά κράτη και από ό,τι καταλαβαίνω, η εισηγήτρια καταλαβαίνει το ειδικό πρόβλημα που αφορά τις ε, βαλτικές χώρες. Μιλάμε για... Δεν μιλάμε ακόμα για το άνοιγμα των αγορών. Θα θέλαμε κι εμείς να μπορέσουμε να ανοίξουμε τη δική μας αγορά, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει έρισμα στην Ευρώπη προς αυτή την κατεύθυνση διότι έχουμε αρχίσει να λειτουργούμε κατά αυτόν τον τρόπο από το 2004 και μετά. Μιλάμε για ένα 35% επιβάρυνσης από τις υποδομές και αν ε, εγκρίνουμε αυτή την πρόταση το χρηματοδοτούμε τρίτες χώρες διότι τα εμπορεύματά μας προέρχονται από τρίτες χώρες κυρίως αυτό, αυτός είναι ένας αγωγός που δεσμεύει τις χώρες οικονομικά και πολιτικά. Χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες λοιπόν, θα ήθελα να πω να δημιουργηθεί μία νέα ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή που να ασχοληθεί με αυτές τις διαφορές, λαμβάνοντας υπόψη και τη διαφορά στους κανόνες, καθώς και διαφοροποίησης, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν ε, διαφορετικές μετρήσεις και υποδομές. Εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε τα ρωσικά πρότυπα. Θα ήθελα λοιπόν να εισακουστούν και οι δικές μας απόψεις. Θα πρέπει να υπάρξουν προσωρινές εξαιρέσεις για αυτές τις χώρες έτσι ώστε η απελευθέρωση να κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο κύριος Μασίνκοβιτς, για τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να λάβετε υπόψη το θέμα των διαμετρημάτων, το, το των σιδηροτροχιών. Νομίζω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε που υπάρχουν διαφοροποιήσεις, τεχνικές διαφοροποιήσεις ως προς το εύρος των σιδηροτροχιών. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Δηλαδή μιλάμε για 1400 χιλιοστά με μία μικρή απόκληση. Άρα, εάν υπάρχει άλλο πάχος, άλλο εύρος, τότε θα υπάρχουν διαφορές και δεν θα μπορούμε να ανταποκριθούμε, όπως ορίζουν και τα κεφάλαια 2 και 3. Ως προς τις, προς τις περιφερειακές υποδομές, πολλές φορές μπορεί να έχουμε ε, διαφορετικά συστήματα εύρους σιδηροτροχιών και γι' αυτό θα πρέπει να μας σε αυτό το θέμα μέσα στα πλαίσια των ε, υποδομών. Εδώ θα πρέπει να μειωθούν τα όρια έτσι ώστε να δώσουμε κίνητρα στους οικονομικούς φορείς και επιχειρηματίες έτσι ώστε να αναπτύξουν το, το δίκτυό τους με νέα συστήματα διαχείρισης. Επίσης, το θέμα είναι κατά πόσο μέσα στα πλαίσια της αδειοδότησης οι οικονομικοί φορείς θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο. Εδώ ε, θα χρειάζονταν επιπρόσθετα κριτήρια για να υπάρξει σύμπτωση. Ο κύριος Κάντσεν για τρία λεπτά. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Πιστεύω ότι μιλάμε για έναν ευρωπαϊκό ενιαίο χώρο των σιδηροδρόμων που θα πρέπει να είναι δελεαστικός και ανταγωνιστικός για να βοηθήσει στη σύσταση του ευρωπαϊκού ενιαίου χώρου. Θα ήθελα να σταθώ σε τρία σημεία. Το πρώτο αφορά την απελευθέρωση του τομέα. Νομίζω ότι θα πρέπει να καλύψουμε αυτό το νομικό κενό. Η μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών έχει ε, απελευθερωθεί, αλλά όχι με μεγάλη επιτυχία. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη αυτή τη μεγάλη ποσοστιαία αναλογία, 70-80% του τομέα όσον αφορά τη μεταφορά επιβατών. Γι' αυτό και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες από το πολιτικό κατεστημένο. Και η εισηγήτρια ενισχύει το ρόλο της Κομισιόν, αν και απότερο στόχος είναι ένας Ευρωπαίος, μια Ευρωπαϊκή ε, Ρυθμιστική Αρχή. Θα πρέπει όλοι οι οικονομικοί φορείς να, μπορέσει, να μπορέσουν να συμμετέχουν σε όλη τη διαδικασία μεταφοράς στους σταθμούς, στη μεταφορά εμπορευμάτων και ούτω καθεξής. Γι' αυτό, επειδή μιλάμε για ιδιωτικοποίηση, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα πρέπει να σταθούμε σε ιδιωτικοποίηση ή απελευθέρωση του τομέα. Θα πρέπει να έχουμε ένα άνοιγμα λοιπόν της αγοράς για τους οικονομικούς φορείς. Αυτό δεν αφορά ένα ενιαίο πρότυπο για τα 27 κράτη-μέλη. Κατανοώ βεβαίως ότι δεν υπάρχει πάντα ενιαίος χαρακτήρας γιατί θα πρέπει να εξασφαλιστεί αυτός ο τομέας και με την εισαγωγή του, των ιδιωτών του ιδιωτικού τομέα. Όσο το τομέας παραμένει κρατικός, μπορεί να υπάρχει ενιαίος χαρακτήρας. Αλλά όταν μιλάμε για διαφοροποίησης και για ιδιωτικοποίηση, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε αυτή την οδό. Δηλαδή το unbundling είναι απολύτως αναγκαίο. Ευχαριστούμε τον κύριο Κάντσον. Μπάτζ τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τα συγχαρητήρια προς την ε, εισηγήτρια. Όλοι ενδιαφέρονται να υπάρξει ένα λειτουργικό σιδηροδρομικό σύστημα που να ικανοποιεί τους ε, επιβάτες, λέει η κυρία ε, Σερακιάνη και εγώ προσθέτω και που να διασφαλίζει καλής ποιότητας θέσεις απασχόλησης. Διαπιστώνω δυστυχώς ότι για άλλη μια φορά όλο το βάρος ρίχνεται στην ανταγωνιστικότητα και πολύ σημαντικά θέματα όπως η διαλειτουργικότητα, δηλαδή η τεχνική εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και άλλα σημαντικά θέματα της χρηματοδότησης των υποδομών των επενδύσεων κατά τη γνώμη μου δεν λαμβάνονται παρκώς υπόψη στο κείμενο της. Για την ρυθμιστική αρχή προσοχή, μην κάνουμε το δεύτερο βήμα πριν από το πρώτο, δηλαδή ναι με να ενισχυθούν τα μέσα που θα διαθέτει η ρυθμιστική αρχή αλλά αυτή θα πρέπει να παραμείνει διαιτητικού χαρακτήρα και όχι να μπορεί να παρεμβαίνει εκ των προτέρων, να μπορεί να παρεμβαίνει μόνο εκ των υστέρων. Ουδής επιθυμεί να αποκλείσει νέους ανταγωνιστές. Η προτινόμενη λύση μου φαίνεται ότι για το λεγόμενο unbundling ότι παρεμβαίνει υπερβολικά στο δικαίωμα κυριότητας και ότι οδηγεί σε μεγάλη γραφειοκρατική επιβάρυνση. η διεθνοποίηση των εξωτερικών στοιχείων κόστους θα οδηγήσει και πάλι σε στρέβλωση του ανταγωνισμού σε βάρος του σιδηροδρόμου. Αργότερα θα μιλήσουμε για την Ευρωβινιέτα. Για τον σιδηρόδρομο εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να είναι δεσμευτικό, δηλαδή το κόστος για το θόρυβο κλπ. θα πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά για το λεγόμενο unbundling και αντίθετα με τον συνάδελφό μου κύριο Ρικέ που μίλησε για εγωισμό των χωρών μελών εγώ θα έλεγα ότι το θέμα αυτό στις χώρες μέλη οι οποίες έχουν συμμορφωθεί με τον νόμο έχουν δηλαδή προβεί σε αναδιαρθρώσεις των ε, ρυθμίσεών τους δεν θα πρέπει να επανέλθουμε και να ζητήσουμε νέες αναδιαρθρώσεις διότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να αναδιαρθρώνονται επάπειρον χωρίς κίνδυνο να καταστραφούν. Θα πρέπει να βασιστούμε σε κοινά μοντέλα, σε, κοινού, σε κοινά πρότυπα, αρκεί να μην υπάρχουν διακρίσεις και πάνω σε αυτά μπορούν να βασιστούν οι ρυθμιστικές αρχές για την ίδρυσή τους. Ερτούκ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική της εργασία που γνωρίζω πόσο δύσκολη ήταν. Δεν θα επαναλάβω πολλά από τα όσα ήδη λέχθηκαν. Θα υπενθυμίσω μόνο λίγα πράγματα. Η κατάσταση όπως παρουσιάζεται σήμερα και γιατί συζητούμε άλλωστε σήμερα οφείλεται σε παραλήψεις της Κομισιόν η οποία δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει ορθή εφαρμογή του πρώτου σιδηροδρομικού πακέτου. Και γι' αυτό ερχόμαστε τώρα να συζητήσουμε αυτό το recast, την αναδιατύπωση. Ας μην το λησμονούμε αυτό. Να μην φορτώνουμε την ευθύνη αλλού. Τα όσα εγκρίνονται στο νομοθετικό επίπεδο πρέπει και να εφαρμόζονται. Δεν μου αρκεί το σχόλιο αυτό. Επιθυμώ να έρθω και σε δύο ακόμη σημαντικά θέματα αφενός την τροπολογία μου 36 για τις υπηρεσίες όπου ο πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτείνεται ότι εάν δεν χρησιμοποιούνται κάποιες υποδομές προσφοράς υπηρεσιών για δύο χρόνια να προωθούνται σε leasing, μακρού χρόνου μίσθωση δηλαδή, ή πώληση εγώ εδώ θέλω να πω ότι είναι σωστό να υπάρχει και το ενδεχόμενο της πώληση, αλλά προτιμώ τα δύο χρόνια και όχι το ένα έτος μόνο που είναι πάρα πολύ σύντομο. Και ένα θέμα ακόμη που δεν θα πρέπει να λησμονηθεί τροπολογία 54 επί του άρθρου 21 στο κείμενο λέει για πιστοποιητικά ασφαλείας της υδρομικής επιχείρησης και όλων των σχετικών και τονίζω εδώ ότι στον τομέα αυτό πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσον οι προδιαγραφές ασφαλείας είναι αρκετά υψηλές. Διότι σε περιοχές της Ευρώπης, σε τμήματα της Ευρώπης, χορηγούνται άδειες ε, οδηγού, ε, μηχανοδηγού στους δρόμου σε πρόσωπα τα οποία δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Ευχαριστώ κυρία Τσικάου. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της. Είναι εξαιρετική αυτή η έκθεση. Θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένα στοιχεία που θεωρώ πολύ σημαντικά. Καταρχήν αναφέρομαι στην ανάγκη συνεχών επενδύσεων στις υποδομές των σιδηροδρόμων, Η έλλειψη επενδύσεων, ακόμα και εκεί όπου έγινε απελευθέρωση, είναι, αποτελεί ένα από τα απότοκα της κρίσης αυτής. Δηλαδή, δυστυχώς δεν έχουν γίνει επενδύσεις, ιδιαίτερα στην συντήρηση των σιδηροδρόμων Γι' αυτό έχουν, έχει πέσει και η ποιότητα των σιδηροδρόμων. Και γι' αυτό ακριβώς οι επιβάτες προτιμούν τη μεταφορά με άλλα μέσα. Η έλλειψη επενδύσεων οδηγεί και σε μείωση του προσωπικού και ένα μεγαλύτερο κίνδυνο ατυχημάτων. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε τις υπηρεσίες και τις συνθήκες εργασίας που να μην πληγούν από την απελευθέρωση και να δούμε και την πραγματική ουσία της διατροπικότητας. Δηλαδή ένας επιβάτης που θέλει να πάει από το σημείο Α στο Β δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσει μια κατάσταση όπου δεν μπορεί να αγοράσει το εισιτήριό του από το σημείο α στο γ, διότι ο οικονομικός φορέας του παρέχει υπηρεσίες μόνο από το σημείο α στο β και όχι από το β στο γ. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η διαλειτουργικότητα. Επίσης πιστεύω ότι και οι σιδηροδρομικές εταιρείες έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση και δεν χρησιμοποιήθηκε το Ταμείο Αντιμετώπισης των Αναγκών για την αντιμετώπιση της παγκοσμιοποίησης. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε τις ανάγκες και της βιομηχανίας και των συνδικάτων. Να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον των συνθήκων εργασίας στο τομέα και να χρησιμοποιήσουμε και αυτό το Ταμείο Αντιμετώπισης της Παγκοσμιοποίησης. Ευχαριστούμε, Ντουράν, τρία λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για την δουλειά της. Την ευχαριστώ και των προτέρων και για τη δουλειά που μένει να κάνει. Θα αναφερθώ στα εξή σημεία. Πρώτα απ' όλα, όπως είπε και ο συνάδελφος Κράμερ, και εγώ πιστεύω ότι τα θετικά από, την, ε, από τον ανταγωνισμό στους σιδηροδρόμους είναι κάτι σχετικό. Μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές τα πλεονεκτήματα αυτά απορροφούνται από τους μεγάλους παίκτε Εκεί που ο κερδίζει ο σιδηρόδρομος από τις οδικές ε, μεταφορές είναι κάτι που οφείλεται και σε άλλους λόγους. Ο διαχωρισμός δεν αποτελεί και εγγύηση, ο κάθετος διαχωρισμός απαραίτητα. Αν θέλουμε μια ε, ενότητα και μια εναρμόνιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν βασικές αρχές, ε, να είναι ακριβείς οι σιδηρόδρομοι, και να δεχτούμε και την ιδέα να έχουμε διαφορετικά μοντέλα και όχι ένα ενιαίο μοντέλο. Να τα δούμε όλα, ανά υπηρεσία, ανά λειτουργία, ποιες, ποια είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία μπορούν να διαχωριστούν και ποια είναι εκείνα που δεν πρέπει να διαχειριστούν για να έχουμε ένα καλό συντονισμό και όχι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σιδηρόδρομοι που έχουν εφαρμόσει τον απόλυτο διαχωρισμό. Έπειτα, οι υπηρεσίες τον έχουμε μια εξωτερική υπηρεσία ενώ ο κορεσμός είναι βασικό στοιχείο, ας προσέξουμε να πρέπει να αποφασίσει μια επιχείρηση για το αν θα είναι διαθέσιμες κάποιες υπηρεσίες που δεν διαθέτει ο ίδιος, αυτό το βρίσκω σαν να πηγαίνουμε υπερβολικά μακριά. Αυτό πιστεύω για την πρόταση Επιτροπής. Για τη χρηματοδότηση τώρα και τις συνθήκες χρηματοδότησης των υποδομών. Καταλαβαίνω τη βούληση της Επιτροπής να βάλει κάποια όρια στα τέλη που θα απαιτήσουν από τις συνδρομικές εταιρείε έτσι κι αλλιώς υπάρχουν μονοπόλια de facto, πρέπει όμως να διασφαλίσουμε σε αυτούς που διαχειρίζονται τις υποδομές τα μέσα ώστε να χρηματοδοτούν και την ανάπτυξη και τη συντήρηση των υποδομών. Και τα κράτη-μέλη πολλές φορές δεν θέλουν ή δεν είναι σε θέση να καλύψουν το κόστος τη διαφορά του κόστους δηλαδή με αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τέλος δεν ξέρω αν το άκουσα εγώ μου το είπανε πάντως το δικαίωμα της απεργίας. Είναι δικαίωμα που υπάρχει και που πρέπει να γίνεται σεβαστό. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μπορούμε να δουλεύουμε με απεργίες που έχουν ε, αναγγελθεί εκ των προτέρων. Και να μπορούμε και να σε αποφύγουμε βέβαια. Μακάρι. Είμαστε σε μια ιδεολογία που θέλουμε ισορροπία. Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι και ενιαίες, αλλά από την άλλη μεριά να μπορούμε να επιτρέψουμε και τον, την ελευθέρωση εκεί όπου αυτό γίνεται. Ο κύριος Πασκορέλη, τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, φοβούμαι ότι θα με αποκεφαλίσετε ως προς το χρόνο εργασίας, διότι δεν θα μπορέσω να αρκεστώ στα τρία έως πέντε λεπτά για να μπορέσω να απαντήσω σε, όλες τις σε όλα τα ενδιαφέροντα σχόλια. Θα κάνετε ό,τι μπορείτε κύριε Πασκουαρέλη, είμαι σίγουρο γι' αυτό. Θα ήθελα να πω ότι η πρώτη ευθύνη της Κομισιόν είναι να εξασφαλίσει τη σιδηροδρομική, την επάρκεια των σιδηροδρόμων με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία κατά τον ε, πιο αποδοτικό τρόπο. Από τη μία πλευρά λοιπόν μας ενδιαφέρουν η καταπαράβαση διαδικασία για να καταπολεμήσουμε την κακή εφαρμογή του πρώτου πακέτου στα κράτη-μέλη και ε, δεύτερον η αναδιατύπωση για να ενισχύσουμε και να εξυγχρονίσουμε το νομοθετικό πακέτο. Υπ' αυτή την έννοια έχουμε προτείνει ορισμένες ε, Διαφοροποιήσεις, χρηματοδότηση, πρόσβαση στις υπηρεσίες και ρόλος και εξουσίες του ρυθμιστή. Η Κομισιόν έχει εκφράσει τη θέση της σε σχέση με την αναδιατύπωση στις ε, δύο προγενέστερες συνεδριάσεις της ΤΡΑΝ, άρα δεν θα επεκταθώ. Θα ήθελα να σχολιάσω ορισμένες τροπολογίες της κυρίας Σερακιάνη, την οποία ευχαριστούμε για την εις εργασία και την ιδιαίτερα ποιοτική εργασία. Θα ήθελα να πω ότι οι τροπολογίες κινούνται προς την κατεύθυνση της πρότασης της Κομισιόν, άρα μπορεί να τις δεχτεί ομαδοποιώντας τις σε σχέση με τις υποδομές, την χρηματοδότηση και τους γενικούς κανόνες για τα ETCS, για τους σύρμους με χαμηλότερη χορύπανση. Όλα αυτά θα τα δούμε στη δεύτερη ανάγνωση. Ως προς τον ρυθμιστή, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν πολλές τροπολογίες για την επανασυστηματοποίηση του θέματος. Δεν θεωρούμε ότι πρόκειται για μια ουσιαστική, για ουσιαστική εργασία, αλλά δεν αντιτάσσεται. Ως προς τη συνεργασία των Ευρωπαίων ρυθμιστών, και του ενιαίου ρυθμιστή. Η τροπολογία 83, οι τροπολογίες 83 έως 88 αποτελούν την κατάλληλη αντιμετώπιση, διότι υπό, την, υπό τις παρούσες συνθήκες δεν μπορούμε εν μία νυχτή να ορίσουμε έναν ενιαίο Ευρωπαίο ρυθμιστή. Η πρόταση Τρεμόζα είναι άκρος ενδιαφέρουσα, αλλά νομίζω ότι οι δημοσιονομικές αρχές θα πρέπει να μας δώσουν πόρους για τους 50 ή 100 νέους υπαλλήλους για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Τόσους χρειαζόμαστε. Ως προς τον συντονισμό μεταξύ Ευρωπαίων ρυθμιστών θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη έναν καλύτερο συντονισμό για τους ε, διαδρόμους, ιδιαίτερα διαδρόμους ε, εμπορευμάτων. Και επίσης οι ρυθμιστές θα πρέπει να είναι σε θέση να επαληθεύσουν τις εργασίες αυτές μέσα στα πλαίσια μιας ευρωπαϊκής ε, ρύθμισης δικτύων. Υπάρχει ένα τρίτο θέμα που μας ανησυχεί ιδιαίτερα ως προς τη ρύθμιση. Ιδιαίτερα αφού άκουσα τις εκκλήσεις των Ευρωβουλευτών για την ανάγκη ενός, ε, μιας ανεξάρτητης αρχής ρύθμισης που να μπορεί να λαμβάνει τάχιστα αποφάσεις. Η τροπολογία 82 μιλά για την ανάκληση. Και αυτός, αυτή η τροπολογία αντιτίθεται με τις αρχές μας, διότι αν θέλουμε μία ανταγωνιστική αρχή, όπως είμαι και πολλοί βουλευτές, θα πρέπει οι αποφάσεις του ρυθμιστικού φορέα να εφαρμόζονται τάχιστα. Προβλέπεται στην πρότασή μας μία ρύθμιση, ε, μία διαμόρφωση αυτού του κανόνα. Δηλαδή, όταν υπάρχει κίνδυνος άμεσης ζημίας ή άμεσης βλάβης, τότε υπάρχει αναστολή, τότε και μόνον τότε υπάρχει αναστολή. Ορισμένοι εκπρόσωποι των βαλτικών χωρών και της Πολωνίας έθεσαν το θέμα των ναύλων ή των υποδομών, της διαφοροποίησης ναύλων. Καταλαβαίνω αυτή τη συλλογιστική, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει ε, θέμα διαφοροποίησης ε, ως προς τους ναύλους. Γνωρίζουμε το πρόβλημα, προσπαθούμε και ε, αναζητούμε μία λύση. Χρειάζεται μεγαλύτερη, χρειάζονται μεγαλύτερες επεξηγήσεις, διότι αυτά τα θέματα έχουν επιληθεί εν μέρη με το παρόν κείμενο, τα προβλήματα που αποσχολούσαν τις βαλτικές χώρες. Μπορώ να σας δώσω και άλλες πληροφορίες διμερώς, αν θέλετε, ως προς τις ε, αδειοδοτήσεις και την ασφάλιση. Θα ήθελα να σας επισύρω την προσοχή στην τροπολογία 54 που ζητεί ώστε η αδειοδότηση που ορίζεται με βάση τις τεχνικές και οικονομικές παραμέτρους να ε, διαθέτει να αφορά και να προϋποθέτει ένα πιστοποιητικό ασφάλειας για τη λειτουργία. Αλλά εάν για την αδειοδότηση προϋποτίθεται το πιστοποιητικό ασφάλειας, με βάση το δίκτυο λειτουργίας αποτελεί πρόσκομα για την ε, εισδοχή στην αγορά. Γιατί πολλά δίκτυα δεν θα υπήρχαν, δεν θα είχαν πρόσβαση στην αγορά εάν είχε εισαχθεί αυτός ο κανόνας στην ε, υπάρχουσα νομοθεσία. Άρα αντιτιθέμεθα. Ως προς την τροπολογία 55 μιλάμε για 100 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος και ανατύχημα. Αυτή είναι η μέγιστη κάλυψη που προϋποτίθεται. Εμείς προσπαθήσαμε να ε, υπαγάγουμε αυτή τη μέγιστη κάλυψη στις προαπαιτήσεις των δικτύων. Όμως υπάρχει μεγάλη ετερογένεια καταστάσεων που αφορούν τα κράτη-μέλη. Άρα 100 εκατομμύρια ευρώ αναέτος και ανατύχημα είναι υπερβολικό. Μιλάμε βεβαίως για μέγιστη κάλυψη, αλλά και πάλι είναι υπερβολικό. Υπάρχει ανάγκη κάλυψης, αλλά νομίζω ότι δεν θα πρέπει να έχουμε ένα τόσο ε, υψηλό όριο, γιατί και αυτό αποτελεί πρόσκομα. Ως προς το unbundling, την αποδέσμευση, θα ήθελα να σας πω ότι η πλήρης θεσμική αποδέσμευση μεταξύ διαχειριστού και επιχείρησης αποτελεί τον πιο απλό τρόπο για να μην έχουμε σύγκρουση συμφερόντων για την ε, απελευθέρωση και την ανταγωνιστικότητα. Το πρώτο ε, πακέτο προέβλεπε κάτι το διαφορετικό. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει σωστή εφαρμογή. Σύμφωνα με την αναδιατύπωση τώρα, δεν θέλουμε να καινοτομήσουμε σε αυτό το θέμα, όμως η Επιτροπή είτε στην αναδιατύπωση είτε στη Λευκή Βίβλο όρισε ότι το 2012 θα προβάλλει μία νέα διατύπωση, μία νέα διάρθρωση που θα οδηγήσει στην πλήρη αποδέσμευση. Για να φτάσουμε όμως σε αυτό και να φτάσουμε και, για και στην ε, απελευθέρωση της αγοράς για τους επιβάτες, χρειάζεται να στεφτεί από επιτυχία αυτή η αναδιατύπωση. Ως προς το δικαίωμα στην απεργία. Δεν θα ήθελα να ε, γίνει κάποια παρεξήγηση εδώ. Κανένας δεν αμφισβητεί το δικαίωμα στην απεργία. Απλώς λέμε σε ένα άρθρο που αποτελεί αντικείμενο τροπολογίας και που αφορά τις συμβάσεις αορίστου χρόνου, ότι θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες διαχείρισης σε περιπτώσεις ε, εξαιρετικής ανάγκης, έκτακτες περιστάσεις. Και αν το προβλέπει η εθνική νομοθεσία μπορεί να προβλέπεται μία ελάχιστη παροχή υπηρεσιών. Το αφήνουμε όμως στο κράτο μέλος, δηλαδή θα δει το κάθε κράτος μέχρι που θέλει να ρυθμίσει. Το τελευταίο θέμα που θέλω να θίξω αφορά τις κατεξουσιοδότηση πράξης. Οι πράξεις αυτές αποτελούν αντικείμενο του ενός ε, τρίτου των τροπολιών Σερακίν. Η συνθήκη είναι σαφής. Το άρθρο 290 μιλά για εξουσιοδότηση, πράξεις κατεξουσιοδότηση όταν πρόκειται για τροποποίηση μη ουσιοδών στοιχείων του κειμένου. Εμείς στις περι... περισσότερες περιπτώσεις, εκεί που ζητούμε αυτές τις πράξεις, το κάνουμε διότι η παλαιά επιτροπολογία με κοινοβουλευτικό έλεγχο έχει μετατρεπεί σε κατεξουσιοδότηση πράξης. Και γι' αυτό απαιτούνται μη ουσιώδεις τροποποίησεις του κειμένου. Υπάρχουν ορισμένε νέες περιπτώσεις όπου ζητούμε κατεξουσιοδότηση πράξης, αλλά αφορούν στοιχεία τα οποία δεν είναι ουσιώδους τύπου το να περιορίσουμε τις πράξεις όπως κάνει η έκθεση προδικάζει το κείμενο αρνητικά και δεν μας επιτρέπει να λαμβάνουμε τάχιστα αποφάσεις για λόγους διαχείρισης. Το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να συναποφασίζει σε τεχνικά και ε, δευτερευούση σημασίας θέματα για την διαχείριση της αγοράς. Ιδιαίτερα ως προς αυτές τις υπηρεσίες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Πριν δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, να προσθέσω κι εγώ κάποια πράγματα. Και θα ξεκινήσω με το στοιχείο κλειδί που είναι το δικαίωμα στην απεργία. Για μένα είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Και ο νόμος αναφέρεται στο πώς λαμβάνεται η απόφαση αυτή, αν υπάρχει κοινοποίηση κτλ. Εντάξει, αλλά δεν θα ήθελε ένα κράτος μέλος να λέει ποιες θα είναι οι ελάχιστες υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρονται στην χώρα μου, για παράδειγμα, μακριά που εκεί που μένω εγώ θα παίρνονται αυτές οι αποφάσεις σε αυτή την περίπτωση και που ξέρουν αυτοί τι θέλω εγώ γιατί χρειάζεται να είναι ελάχιστες υπηρεσίες. Λοιπόν, εγώ λέω ότι υπάρχει το δικαίωμα να αποσύρονται οι εργαζόμενοι. Αυτό είναι το δικαίωμα βασικά. Είναι η εθνική διάσταση που μπαίνει εδώ πολύ. Και τελικά, ποιος θα αποφασίσει τι θα κάνουν οι σιδηρόδρομοι και περί τίνος πρόκειται. Υπάρχει η δυνατότητα εδώ πέρα εισόδου στην αγορά. Αυτό είναι στοιχείο κλειδί. Πρέπει να υπάρχουν ε, ίδιες προϋποθέσεις για όλους τους σιδηροδρόμους στην Ευρώπη και για μένα για καιρό υπήρχαν κυρίαρχες δυνάμεις στην Ευρώπη που καθόριζαν το τι θα γίνεται στην αγορά αυτή. Το θέμα της διαλειτουργικότητας επίσης είναι σημαντικό. Πρέπει να έχουμε ένα τέτοιο δίκτυο γιατί μόνο τότε θα είναι ανταγωνιστικό το σιδηροδρομικό μας δίκτυο, ανταγωνιστικό ως προς τις οδικές μεταφορές. Έρχομαι και στην αποσύνδεση, το unbundling τι θέλουμε, θέλουμε έτσι όπως είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο με την ιδιωτικοποίηση. Εγώ δεν θα ήθελα κάτι τέτοιο, είναι μια σκέτη καταστροφή. Άσε που και πτώχευση. Και το κράτος τελικά πλήρωσε περισσότερα από τα χρήματα των φορολογούμενων για, τις, για τους ιδιωτικοποιημένους σιδηροδρόμους από ό,τι πλήρωνε πριν για τους κρατικούς σιδηροδρόμους. Εδώ λέμε ότι ο φορέας είναι κάτι σαν ε, βοηθός του κύριου φορέα. Όχι, πρέπει να υπάρχει ανεξαρτησία και πρέπει να υπάρχει ο διαχωρισμός κάπου. Είτε το ονομάζετε unbundling, είτε το ονομάζετε κάπως αλλιώς, δεν με νοιάζει εμένα. Αλλά μέσα σε μια ανταγωνιστική αγορά δεν μπορούμε να έχουμε ένα διαχειριστή υποδομών ο οποίος να βρίσκεται στη διαγραφή και πληρώνεται από ε, τους ίδιους. Και έρχομαι και στο τελευταίο. Πολλά κράτη-μέλη το έχουν σημειώσει και είναι το θέμα του ρυθμιστή. Κάποιοι από τους ρυθμιστές δεν κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει. Γιατί τελικά δεν λειτουργούν ως ρυθμιστές τα κράτη-μέλη πρέπει να κοιτάξουν προσεκτικά και να δούνε τελικά τι λένε ότι ισχύει για τον ρυθμιστή των σιδηροδρόμων. Χρειάζεται ένας ανεξάρτητος ρυθμιστής που να δράμε διαφάνεια, απόλυτη, ώστε όλοι να μπορούν να δουν τι ακριβώς γίνεται. Γιατί ο ρυθμιστής είναι εκεί για να ρυθμίσει τους σιδηροδρόμους και όχι για να ευνοεί το ένα ή το άλλο τμήμα των σιδηροδρόμων. Άρα τα στοιχεία κλειδί αυτά πρέπει να τα προωθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο με τις τροπολογίες μας. Γιατί τελικά αυτό που θέλουμε όλοι είναι να πετύχουν οι σιδηροδρόμοι. Όλοι αυτό λέμε, ότι θέλουμε οι σιδηρόδρομοι να πετύχουν. Αλλά μην υποτιμάτε τη δυνατότητα των σιδηροδρόμων να σας προσφέρουν περισσότερους λόγους για να μην το κάνετε παρά για να το κάνετε. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να θέσουμε το πλαίσιο έτσι ώστε να υπάρξει πρόοδος στους σιδηροδρόμους. Εξάλλου, μερικοί από εμά αναγκάζονται να καταπιούν το χάπι της εθνικής περηφάνειας και να δούνε τα πράγματα από ευρωπαϊκή οπτική γωνία και όχι από εθνική οπτική γωνία. Η κυρία Σαρακιάνη τώρα, τι έχετε να προσθέσετε. Ευχαριστώ. Απλώς θα ήθελα να κάνω ορισμένες διασαφήσεις. Βεβαίως γνωρίζω ότι έχω πολύ λίγο χρόνο στη διαθέσή μου. Θα έρθω σε επαφή με τους συναδέλφους και θα μιλήσουμε για λεπτομέρειες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μπράιαν, χωρίς τον οποίο δεν θα είχα το θάρρος να συντάξω αυτή την γνωμοδότηση. Γι' αυτό τον ευχαριστώ για την υποστήριξή του Συμφωνώ με τον κύριο Κούν όταν ε, μιλά για τη διαφάνεια που είναι το κλειδί της αναδιατύπωσης, στην διαχείριση στους λογαριασμούς, στις υποδομές γενικότερα και γνωρίζω ότι η ενδιαφέρουσα σημερινή συζήτηση και σας ευχαριστώ όλους για το ότι συνεισφέρατε εις βάθος. Θα ήθελα λοιπόν, λοιπόν ότι όλη αυτή η κατάσταση είναι το πολιτικών αποφάσεων που θα πρέπει να ληφθούν. Και ενώ κατανοώ αυτά που είπε ο κύριος Τρεμόζα, δεν συμφωνώ με αυτόν όταν είπε ότι θα πρέπει να αναμείνουμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Γνωρίζουμε ότι το πρώτο πακέτο απέτυχε, ξέρουμε ότι θα πρέπει να αναδιατυπωθεί και δεν θα το κάνει αυτό το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς φέρουμε την πολιτική ευθύνη της ε, πλήρους αναδιατύπωσης. Δεν ασχολήθηκε υπερβολικά με την αποδέσμευση. Αν δείτε το κείμενο της έκθεσης μου, λιγότερα από 10 άρθρα ασχολούνται με την αποδέσμευση και 110 είναι τα συνολικά άρθρα. Δηλαδή ε, ασχολήθηκα επαρκώς αλλά όχι υπερβολικά. Εάν υπήρχε μια σαφής πρόταση από την Κομισιόν που θα μας ορίσει αυτό το διαχωρισμό επακριβώς και με βάση τη Λευκή Βίβλο, ίσως τώρα θα ήταν εύκολα από πολιτικής άποψης να φτάσουμε σε μια συμφωνία αναλαμβάνοντας το πολιτικό κόστος αυτών των αποφάσεων. Επίσης, νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ιδιαιτερότητα ορισμένων χωρών. Ε, με τον κύριο Τζίλερ ε, ασχολήθηκα δηλαδή με τις βαλτικές χώρες και θα ήθελα να συνεργαστούμε για να εξεύρουμε την καλύτερη δυνατή λύση, διότι αυτές οι χώρες διαφέρουν ανάλογα με το σιδηροδρομικό σύστημα που ισχύει. Ως προς την ασφάλιση, αυτό που προβλέπετε στην τροπολογία 55 δεν είναι η μέγιστη κάλυψη αλλά η ελάχιστη. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να δούμε κατά πόσο έχει μεταφραστεί σωστά διότι έγινε λόγος για μέγιστη κάλυψη ενώ είναι ελάχιστη η κάλυψη που προβλέπεται στην τροπολογία 55 ως προς το δικαίωμα για απεργία και εγώ συμφωνώ ότι δεν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την αρχική πρόταση της Κομισιόν. Πρόβαλα μία τροποποίηση, αλλά επειδή πολλά κράτη έχουν διατάξεις συνταγματικού χαρακτήρα που ορίζουν το δικαίωμα στην απεργία, δεν χρειάστηκε ε, να υπησέλθω σε αυτό το θέμα, γιατί θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγχυση. Βεβαίως, ως προς την αρχή της τροποποίησης της αρχικής πρόταση της Επιτροπής ε, συμφωνώ ως προς τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξης θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ε, ορίσει αυτές τις αρχές έχουν αλλάξει ορισμένα θέματα που υπάρχουν στις, ε, εντάσσονται στις κατεξουδότηση πράξης. Η δική μου προσέγγιση αφορά την θέληση πολλών συναδέλφων να ενισχύσουμε την αρχή του ρυθμιστή, της ρυθμιστικής αρχής και θα ήθελα να μου κάνετε υποδείξεις για αυτή την ενίσχυση ως προς το πρόσωπα του Ευρωπαίου ρυθμιστή και εδώ έχω υποβάλει τροπολογίες διότι εδώ υπάρχει ένα νομικό κενό και δεν μπορεί να ενταχθεί στην πρόταση οδηγίας στα πλαίσια της αναδιο... αναδιατύπωσης ως προς τις αδειοδοτήσεις νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να φτάσουμε στην ευρωπαϊκή άδεια. Ίσως θα μπορούσαμε να προβάλλουμε συγκεκριμένες πολιτικές δεσμεύσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, σε σχέση με την δυνατότητα μεταφοράς στις, ε, στον εθνικό τομέα, ως προς τις εθνικές μεταφορές, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτή η παρέκταση. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Γκρός που δέχτηκε αυτή την ε, πρόκληση εγώ δεν εφήβρα τίποτα το καινούριο, απλώς εφαρμόζω αυτά που προϋπάρχουν. Σας υπενθυμίζω ότι τον Ιούνιο του 2010 το Κοινοβούλιο ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία ένα ψήφισμα για το άνοιγμα της αγοράς των σιδηροδρόμων με τον διαχωρισμό αυτό και την ανεξαρτησία. Άρα απλώς εφαρμόζουμε αρχές που έχουν προαποφασιστεί για να έχουμε μια ανοιχτή και διαφωνή αγορά η οποία να εγγυάται τις συνθήκες εργασίας και τις κοινωνικές ρήτρε κινητικότητας και εργαζομένων. Πιστεύω ότι μπορούμε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση με σαφείς κανόνες το αγγλικό σύστημα που υπενθύμισε ο Μπράιαν δεν είναι το σύστημα που λαμβάνουμε ως σημείο αναφοράς. Κανένα σύστημα δεν αποτελεί σημείο αναφοράς εδώ. Οικοδομούμε κάτι διαφορετικό με βάση επιμέρους σημεία για να βελτιώσουμε το σιδηροδρομικό σύστημα. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες, σαφείς κανόνες κανόνες διαφάνειας και ανεξαρτησίας καθώς και εποπτείας της αγοράς των σιδηροδρόμων. Ως προς τροπολογία 36, γιατί αναφέρομαι σε ένα χρόνο, διότι το Κοινοβούλιο θέλει να κόψει δύο, τα δύο χρόνια. Θα πρέπει να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε, διότι δεν πρέπει να κολλησιεργούμε. Θα πρέπει να έχουμε το πολιτικό στένος να κάνουμε πολύ περισσότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την εισηγητρία. Ήταν ένα πολύ σημαντικό θέμα, γι' αυτό και τράβηξε τόσο. Και επίσης ήταν πολύ σημαντικό να έχουν πει όλη την γνώμη τους. 30 Μαΐου είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες στη συνάντησή μας του Ιουνίου. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας τον Ιούλιο και στην Ολομέλεια τον Σεπτέμβριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την εισηγήτρια και περνάμε στο επόμενο θέμα μας που είναι η Ευρωβινιέτα. Η εισηγητής είναι ο κύριος Αλκαντραουή και πρόκειται για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, ο κύριος Ελκατράβη να μας πει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω καλά νέα. Βάσει της εντολής που πήρα από την Επιτροπή Μεταφορών στη δεύτερη ανάγνωση και μετά από συνεργασία με τους κοιόδης συζητητές, χθες το βράδυ καταλήξαμε στον τριμερή διάλογο σε κάποια συμφωνία. Βεβαιωμένη να επιβεβαιωθεί τον Ιούνιο στην Ολομέλεια. Πρέπει να σας πω ευθύ αμέσω ότι αντιλαμβάνομαι ότι κανείς δεν θα είναι ευτυχής 100% από την συμφωνία αυτή, αλλά αυτή είναι, αυτό είναι και το νόημα κάθε συμβιβασμού. Προσωπικά λοιπόν εγώ πιστεύω ότι έχουμε μια ισορροπημένη συμφωνία, μια καλή συμφωνία. Βάσει της αρχής ο πληρώνει όσον αφορά τις μεταφορές. Για πρώτη φορά λοιπόν έχουμε αυτή την αρχή για την οποία αγωνιζόμαστε τόσο πολύ καιρό, την εξωτερήκευση του κόστους επίσης, κάτι το οποίο πάντα θέλαμε. Δεν είναι αυτό το τέλος. Είναι όμως ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα μπρος. Εδώ και χρόνια αγωνιζόμαστε. Τώρα θα συνεχίσουμε με την Ευρωβινιέτα να πετύχουμε ακόμα περισσότερα. Μετά δηλαδή την επίτευξη του πνεύματος που θέλαμε να πετύχουμε, από εδώ και πέρα πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα για την επίτευξη και της ουσίας. Τώρα, τι περιλαμβάνει η συμφωνία που πετύχαμε χτες το βράδυ και για την οποία ζητάω κατεστήριξή σας. Πρώτα απ' όλα, αναφέρεται στην, ε, στις υποδομές, ε, στα τέλη, υπάρχει για το θέμα του εξωτερικού κόστους που πετυχαίνουμε επίσης και τέλος υπάρχει και το θέμα της αρχής του ορυπαίνου πληρώνει. Τώρα για το θέμα της, ε, του κόστου συμφόρησης. Αυτό δεν υπολογίζεται ξεχωριστά. Δεν ε, θα υπήρχε έτσι καλλιώς πλειοψηφία ούτε εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά ένα τμήμα περιλαμβάνεται ε, δεδομένου ότι δεχόμαστε πολύ περισσότερους μηχανισμούς διακύμανσης της χρέωσης. Ε, μιλάμε για ανώτατα επίπεδα συμφόρεσης και βάζουμε κάποια ανώτατα όρια. Αυτό θέλει το Συμβούλιο. Εγώ προσωπικά θα προτιμούσαν, είχαμε πάει ακόμα πιο μακριά για να συμπεριλάβουμε και τον αριθμό των ωρών, πέντε ώρες ε, συμφόρηση. Αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχουμε. Κρατήσαμε το θέμα της διακύμανσης που μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη. Αυτό ναι. Και από εκεί και πέρα τίποτα άλλο. Αλλά ήδη αυτό είναι πολύ σημαντικό και όπως σας είπα συμπεριλαμβάνεται και το στοιχείο της συμφόρησης στο μοντέλο αυτό. Κατά τα άλλα, ετέθη ένα θέμα για τους χρήστες. Να είναι πιο απλά τα πράγματα και έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει κάποιο είδους οδηγό για τους χρήστες ώστε να ξέρουν οι χρήστες για την κάθε χώρα τι τέλη επιβάλλει. και πρέπει να ενημερώνεται αυτός ο οδηγός για να ξέρουμε ότι ανταποκρίνεται πάντα στην πραγματικότητα που ισχύει στις διάφορες χώρες. Τώρα για την ε, αγορά. Εμείς θέλαμε να είναι εφικτό να γίνεται διάκριση ανάμεσα στα φορτηγά που είναι πιο καθαρά, που ανταποκρίνονται δηλαδή στις προδιαγραφές ευρώ, ε, και διάκριση με τα άλλα τα πιο παλιά φορτηγά, τα λιγότερο καθαρά, που ρηπαίνουν περισσότερο. Να λαμβάνετε υπόψη δηλαδή και αυτό το στοιχείο και υποδομές και συμφόρηση για τις ε, κατηγορίες ε, που προβλέπουμε και το εξωτερικό κόστος να λαμβάνεται πλήρως υπόψη. Η μεγαλύτερη απέτηση που είχε δικιά μας η Επιτροπή ήταν αυτή που βρίσκουμε και στον συμβιβασμό, δηλαδή μεγάλη δέσμευση από τα κράτη-μέλη, ότι τόσο τα έσοδα όσο και τα τέλη από τις υποδομές και το εξωτερικό κόστος, όλα αυτά τα έσοδα θα χρησιμοποιούνται για καλύτερες μεταφορές, πιο βιώσιμες υποδομές και μεταφορές. 15% τουλάχιστον πρέπει να επενδύεται στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Αυτή την παράγραφο βέβαια πρέπει να τη δούμε μαζί με την παράγραφο που αναφέρεται στη διαφάνεια. Γιατί δεν είναι μόνο σημαντικό τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν τα χρήματα, είναι πολύ βασικό και το κοινό και αυτοί που πληρώνουν, οι φορολογούμενοι, αυτοί που πληρώνουν γενικότερα οι να ξέρουν που πάνε τα χρήματά τους. Και γι' αυτό πετύχαμε κάτι πολύ σημαντικό. Τα κράτη-μέλη αναλαμβάνουν τη δέσμευση σε τακτικά χρονικά διαστήματα να υποβάλουν έκθεση στην οποία να αναφέρεται πού ακριβώς έχουν πάει τα χρήματα. Με κάθε λεπτομέρεια. Τι μεταβολές υπάρχουν στα τέλη, τι διακυμάνσεις και για τα έσοδα από τις υποδομές και ε, από το εξωτερικό κόστος. Τα κράτη-μέλη πρέπει να πείθουν, να δείχνουν πραγματικά πώς χρησιμοποίησαν τα χρήματα και πώς στήρισαν τις δεσμεύσεις τους για τις επενδύσεις που υποχρεούνται να κάνουν από τα έσοδα στις υποδομές και στις μεταφορές. Πρέπει να εξηγούν δηλαδή τι δράσεις ανέλαβαν για να πετύχουν τη δέσμευση αυτή που έχουν αναλάβει. Κάτι άλλο σημαντικό για μας είναι η διαλειτουργικότητα. Ε, δεν θέλουμε να καταλήξουμε με 26 διαφορετικά συστήματα όπου οι οδηγοί των φορτηγών να ε, πρέπει να έχουν ολόκληρο οδηγό για να κυκλοφορούν ε, μέσα στην Ευρώπη. Θέλουμε να υπάρχει ένα σύστημα και μόνο με τον οποίο να μπορούν να κυκλοφορούν μέσα στην Ευρώπη. Για την εφαρμογή τώρα, το γεωγραφικό θέμα δεν ήταν το πιο σημαντικό, παραμένει λίγο πολύ το ίδιο, έχουμε το TEN 10. Αλλά υπάρχουν βέβαια και τα τμήματα εκείνα που δεν περιλαμβάνονται στο ten 10. Το πιο επίμαχο θέμα ήταν το θέμα του βάρους των φορτηγών, της χωρητικότητας. Το Σεβούλιο θέλει κάποια ελαστικότητα εκεί. Ε, μιλούσαν για 12 τόνους και κατέληξαν στους 3,5 τόνους. Τελικά είπαμε ότι προς το παρόν αρχίζουμε από τους 12 τόνους και οι 3,5 τόνοι θα ισχύσουν από το 2013. Και οι 12 τόνοι πόρους. κυρίως όταν μέρος ε, της διαδρομής γίνεται από μικρότερους δρόμους. Αφήσαμε κάπως πιο ελεύθερα τα πράγματα εδώ. Το σημαντικό πάντως είναι ότι τα κράτη-μέλη που θέλουν να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να το ανακοινώνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ξεκινάνε, όπως είπαμε, από τους 12 τόνους. Δύο πράγματα ακόμα. Πρώτο, τα επόμενα βήματα. Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Όπως σας είπα και στην αρχή δεν τελειώνει εδώ η διαδικασία. Εδώ ξεκινάει η διαδικασία της εσωτερήκευσης του εξωτερικού κόστους. Η Ευρωπαϊκή μένει να κάνει πολλή δουλειά ακόμα τα επόμενα χρόνια θα ερευνήσει για να δει τι άλλοι τρόποι μεταφορών μπορούν να συμπεριληφθούν σε αυτό το σύστημα ή πρέπει να προσθεθεί και άλλο εξωτερικό κόστος και άλλα. Τώρα δεν θα σας πω ολόκληρο τον κατάλογο, πάντως θέλουμε να διευρυνθεί η υπόθεση αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να το ψάξει αυτό και να μας ενημερώσει μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια. Και μέσα σε επόμενους μήνες θα υπάρξει μία έκθεση που θα λέει τι μέτρα μπορούν να ληφθούν ακόμα ώστε να υπάρξει εσωτερήκευση του εξωτερικού κόστους και τι μέτρα πρέπει να ακολουθήσουν. Τέλος, τέλος, ένα τεχνικό ζήτημα γίνεται συζήτηση μεταξύ Επιτροπής Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για να εξηγήσουμε στα κράτη-μέλη με ποιο τρόπο πρέπει να εκπονούν την νομοθεσία. Έχουμε βρει μια λύση πριν καταλήξουμε σε κάποια οριστική με μια διευκρίνηση που πρέπει να κάνει το Συμβούλιο μαζί με το Κοινοβούλιο και θα αρκεί για να μην θεωρηθεί ότι υπάρχει προηγούμενο. Αυτά, Πρόεδρε. Προσπάθησα μέσα σε λίγα λεπτά να σας παρουσιάσω την ουσία των όσων πετύχαμε. Η γνώμη μου είναι και η συμβουλή μου να στηρίξουμε την συμφωνία αυτή στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ που είναι μια συμβαστική συμφωνία. Πρόεδρος, ωραία, ευχαριστούμε για την πλήρη αυτή εξήγηση και παρουσίαση. Ο κύριος Δεγρός, πρώτα τρία λεπτά, τρία λεπτά ο καθομιλητής. Ευχαριστώ. Η κυρία Βόρτμαν Κόλ συμμετέχει σε τριμερή διάλογο και γι' αυτό στο όνομά της αλλά και στο όνομα του Λαϊκού Κόμματος θα πω πρώτα ότι ευχαριστούμε τον εισηγητή ότι ειλικρινώς είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα διότι βέβαια δεν είναι και εύκολο σε τέτοιο θέμα για τις περιφέρειες, απομακρυσμένες περιφέρειες, τις ε, μικρές και μεγάλες χώρες μέλη. Όλα αυτά λοιπόν να ενταχθούν σε ένα ενίο κείμενο. Περάσαμε πολύ κοντά από το μηδέν θα έλεγα και ο εισηγητή μπόρεσε και διέσωσε ορισμένα πράγματα και αυτά μας ικανοποιούν. Πράγματα τα οποία προδιετίας φαίνονταν αδύνατον να υλοποιηθούν, τώρα φαίνεται ότι είναι πραγματοποιήσιμα. Για μας η σημαντική ήταν η διαλειτουργικότητα, το earmarking και σε ό,τι αφορά τις παραλλαγές να μην πάμε υπερβολικά προς τα κάτω ή προς τα πάνω. Και νομίζω ότι αυτοί οι τρεις στόχοι επιτυγχάνονται. Ίσως όχι στο βαθμό όπως θα ήλπιζαν ορισμένοι. Η διαλειτουργικότητα για μας φαινόταν κάτι το αυτονόητο, τώρα πάει να γίνει πιο αργά βέβαια. Αυτό το earmarking, ας το πω καλύτερα, mini earmarking, είναι ωστόσο ένα πρώτο βήμα προς μια κατεύθυνση που ε, θα δώσει ανατολισμό και για άλλες υποθέσεις ε, στο μέλλον. Η Ευρω 3 νομίζω αποτελεί εν προκειμένου μια θετική συμβαστική λύση και θα ήταν κρίμα εάν σε σύγκριση με τα όσα ήδη είχαμε πετύχει το 2008 δεν είχαμε επιτύχει γιατί 3,5 τόνους βρίσκω καλό και η δυνατότητα για τα τόνα για ορισμένες χώρες βρίσκω ότι και αυτή είναι σημαντική αλλά νομίζω ότι καλά προσεγγίζουμε τον τομέα. Τελευταίο σχόλιο αυτοί η πίνακες συσχετισμού νομίζω ότι δεν επιτρέπεται να δώσουμε, να φτιάξουμε εδώ ένα ε, προηγούμενο, γιατί και τίποτε άλλο, να δώσουμε ένα καθαρό μήνυμα στο Συμβούλιο. Θέλουμε μια σαφή δήλωση του Συμβουλίου, εάν πρόκειται τώρα για πολύ μικρές τροποποιήσεις, όπως είναι προκειμένο, και κινδυνεύουμε να χάσουμε προθεσμίες λόγω αυτών και να καταλήξουμε σε περιτές ε, διαιτητικές διαδικασίες, τότε καλύτερα το αφήσουμε. Βρίσκω λοιπόν ότι είναι ικανοποιητικό το αποτέλεσμα και ευχαριστώ όλες και όλους όσοι συμμετέσχουν στις εργασίες. Στέρξ, τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Πολύ καλά το είπε ο Ματιέ. Ότι περάσαμε πολύ κοντά από το μηδέν. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω και να ευχηθώ στον εισηγητή. Το θέμα ήταν πώς θα χάσουμε λιγότερα και θα κερδίσουμε περισσότερα είμαστε αδύναμος κρίκος της συμφωνίας. Το earmarking δεν είναι αυτό που θέλαμε. Είπαμε τα κράτη-μέλη shall, member states shall. Για την συμφόρηση ζητήσαμε η ίδια μεταχείριση για όλους. Δεν υπάρχει. Αυτά είναι τα δύναμα σημεία. Το ξέρουμε. Τι κερδίσαμε όμως. Υπάρχει κάτι για το earmarking. Το Συμβούλιο δεν ήθελε τίποτα. Έλεγε ούτε να τα ακούμε. Όμως υπάρχει. Member States should δεν είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που θα θέλαμε εμείς, αλλά κάτι υπάρχει για το earmarking. Ξέρουμε πόσα χρήματα είναι και ποιες είναι οι δράσεις που αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη από τα έσοδα από το εξωτερικό κόστος. Ένα δεύτερο σημαντικό σημείο είναι, όπως είπε και ο Ματιέ, η λειτουργικότητα. και αυτό είναι βασικό στα πλαίσια της εφαρμογής και για την εσωτερική αγορά για μένα είναι πολύ σημαντικό. Αν δεν το είχαμε αυτό, τότε θα είχαν τη διτάση τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν διαφορετικά συστήματα. Τώρα, στρατηγικά αυτό που έχει σημασία είναι να απαγιωθεί αυτή η αρχή. Γιατί συμποθέσουμε υποθέσουμε ότι δεν θα το κάνουν. Μετά έρχονται όλα τα επόμενα σημεία. Και όλα αυτά τα κεφάλαια εξωτερι... μάλλον εσωτερικεύση του εξωτερικού κόστους. Διαφάνεια για άλλες μορφές μεταφορών. Η υποχρεωτική εφαρμογή της ε, Ευρωβινιέτας. Δεν συζητιέται καν. Οπότε, όπως είπες, και το είπα και χτες στον τριμερή διάλογο, είμαστε στην αρχή της συζήτησης. Και μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια θα ξανασυζητήσουμε. Σε δύο χρόνια από τώρα ήδη θα αρχίσουμε. Για τις οδικές μεταφορές, για άλλες μεταφορές, με ποιο τρόπο θα προχωρήσουμε. Η ομάδα μου τουλάχιστον, και το έχω πει και στον εισηγητή και το ξέρω ότι δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα, θα το υποστηρίξω αυτό στην ομάδα μου, ότι υπάρχουν κάποια δύναμα σημεία, λέγω την ε, έκθεση αυτή θα την υποστηρίξω. Τη θέση μας θα την υποστηρίξω στην ομάδα μου. Ε, είσαι ο καλύτερος για να πείσεις τους φιλελεύθερους. Η κυρία Λίχτεμπέργκερ, τρία λεπτά παρακαλώ. Εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξη μετά από αυτό τον τριμερό, τριμερή συγγνώμη, διάλογο. Όποιοι ανέμεναν ότι οι οδικές μεταφορές εμπορευμάτων θα αρχίσουν να κάνουν κάποια πρώτα βήματα προς μια βιωσιμότητα, προς μια αηφορία μάλλον περιβαλλοντική, θα έχει απογοητευτεί. Ο συνάδελφός μας είπε ότι φτάσαμε να αγγίξουμε το μηδέν. Εγώ νομίζω ότι μείναμε κιόλας πολύ κοντά στο μηδέν. Δεν ε, ε, ευθύνεται εδώ δόλος ο εισηγητής, το τονίζω αυτό, ο οποίος κατέβαλε προσπάθειες. Ευθύνεται το γεγονός ότι η σφικοφολιά των λομπιστών, των λόμπι, βρίσκεται στο Συμβούλιο και οι κυβερνήσεις είναι εκείνες οι οποίες δεν θέλουν να κάνουν απολύτως τίποτε για να λάβουν μέτρα που θα ενισχύσουν την αηφορία. Όποιος ενδιαφέρεται δηλαδή για παράδειγμα για την ποιότητα ζωής των προσώπων που κατοικούν κοντά σε αυτοκινητοδρόμους θα δει να του σηκώνονται οι τρίχες να ανατριχιάζει από τα πράγματα που βλέπει. Δηλαδή αύξηση των φορτηγών αυτοκινήτων οι ρυθμίσεις για τον περιορισμό του τονάζ με πίεση μιας από τις μεγαλύτερες χώρες μέλη της Γερμανίας δηλαδή αποδυναμώνονται και πάλι σχετικές διατάξεις διαπιστώνουμε ότι το Συμβούλιο Υπουργών κάθε τι που έχει σχέση με ευρωπαϊκή πολιτική αηφορίας τα φρενάρει. Πρόκειται για διαπίστωση γεγονότος την οποία οφείλουμε να κάνουμε διότι ένα πράγμα είναι σαφές με την μορφή αυτή θα καταστεί πολύ δύσκολο οποιαδήποτε χώρα μέλος να εφαρμόσει οτιδήποτε. Και έτσι πράγματι δεν πετυχαίνουμε και πολλά πράγματα. Δηλαδή η αντιπαράθεση θα διαρκέσει, θα συνεχιστεί και κάτι που πρέπει να σημειώσουμε είναι η απογοήτευση των ανθρώπων εκείνων που ανέμεναν από το ευρωπαϊκό επίπεδο να τηρήσει, να υλοποιήσει αυτά που υπόσχεται με κάθε επίσημη ευκαιρία. Δηλαδή αηφορία στις ε, σεβασμό του περιβάλλοντος στις μεταφορές. Ότι αυτή η ελπίδα τους λοιπόν δεν πληρούνται. Και αυτά βαρύνουν το Συμβούλιο. Και αυτό πρέπει να είναι ο αποδέκτης, το Συμβούλιο δηλαδή, ε, πάσης καταγγελίας και παντός παραπώνου. Ευχαριστώ κύριο Ζήλε. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Η ομάδα μας είναι ικανοποιημένη με αυτό το συμβιβασμό. Όπως γνωρίζετε, δεν έχουμε εισαγάγει άλλες προτάσεις. Γνωρίζουμε πόσο δύσκολο ήταν να συμφωνηθεί αυτό το, από το Συμβούλιο. Θελήσαμε δεύτερη ανάγνωση, αλλά στη, με βάση τη διαδικασία συνδιαλλαγής Ίσως αυτό το αποτέλεσμα. Ο κύριος Αλκαντράουι ε, έχει επιτελέσει εξαιρετική εργασία και η έγκριση αυτής της ε, θέσης είναι πολύ σημαντική. Νομίζω ότι κάτι καταφέραμε εδώ με στοιχεία τα οποία εξέλιπαν στο παρελθόν και νομίζω ότι το θέμα της Ευρωβινιέτας είναι κάτι που μπορεί να ε, χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη μέσα στα πλαίσια της ρήπανσης. Έχουμε ένα ε, ενιαίο τέλος υποδομών. Μερικοί δεν ε, θέλησαν να το θίξουν. Στη Λετωνία, Εστονία και Λιθουανία που χρησιμοποιείται ε, ένα μέρος του ρωσικού δικτύου δεν υπήρξε προθυμία να χρησιμοποιηθεί η Ευρωβινιέτα. Άλλες, και άλλες χώρες είναι επιφυλακτικές διότι δεν υπάρχει πολιτική θέληση δεν θα μπορέσουμε να ε, το κάνουμε αποδεκτό στη χώρα μου στο εγγύς μέλλον. Κανείς δεν είναι ικανοποιημένος με την ε, κατάσταση. Εμείς χρησιμοποιούμε το οδικό ε, δίκτυο, βεβαίως τα βαρέα φορτηγά μολύνουν. Αλλά το θέμα είναι κατά πόσο υπάρχει ε, επαρκής χρηματοδότηση. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι. για τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι ο εισηγητής, ο κύριος Ελκαντράουι, ε, τα κατάφερε πολύ καλά, διότι η εντολή ήταν να υποστηρίξει τη θέση της ε, πλειοψηφίας. Εμείς όμως, ούτε η χώρα μου, ούτε εγώ ανήκουμε στην πλειοψηφία. Είμαστε αντιφρονούντες. Γι' αυτό θα πρέπει να εξαιρεθούμε. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να είμαστε, να σταθούμε πιστοί εμείς περάσαμε από την καταψήφιση στην αποχή. Αυτό είπαμε στην Επιτροπή Μεταφορών την τελευταία φορά και γνωρίζουμε τις μεγάλες δυσκολίες που υπάρχουν, γιατί δεν πρόκειται για ένα θέμα λόμπι. Όμως τα κράτη, ας μην τραπούμε να το πούμε, έχουν διαφορετικά συμφέροντα ανάλογα με το αν ευεργετούνται ή όχι δεν θα πρέπει να μιλήσουμε για αηφορία ή βιωσιμότητα. Μας ενδιαφέρει ποιος πληρώνει και ποιος ε, εισπράττει. Τα ωραία λόγια δεν αρκούν. Νομίζω ότι και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατέβαλαν μια προσπάθεια συνάντησης και τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου οδήγησαν σε μία εξισορρόπηση κατά το δυνατό. Θα μελετήσουμε αυτές τις συμφωνίες εις βάθος. Κύριε Αλκαντράουι, δεν θα μπορέσω δυστυχώς να κινηθώ πέραν αυτού, πέραν αυτής της υποχώρησης, αλλά θα προσπαθήσουμε να δείξουμε κατανόηση γιατί είμαστε μεν αντιφρονούντες, αλλά δεν θα θέλαμε να αποτελέσουμε τροχοπέδι σε μια γενικότερη συμφωνία. Και μετά από μία λεπτομερή μελέτη βλέπουμε, θα δούμε ποια ε, είναι τα συμφέροντα της δικής μου χώρας και άλλων χωρών που είναι περιφερειακές χώρες που ε, θεωρούν ότι η Ευρωβινιέτα είναι πανάκια. Δεν είναι πανάκια. Δεν σας προσάπτω τίποτα κύριε Αλκαντράουι. Εμείς ε, προβαίνουμε σε μία ε, περισυλλογή και προχωρήσαμε πολύ μακριά από την αρχική μας θέση. Ευχαριστώ. Πρώτο, θέλω να πω ειλικρινέστατα συγχαρητήρια στον εισηγητή για τα όσα επέτυχε. Όχι τόσο για το ουσιαστικό περιεχόμενο, αυτό το συζητούμε, αλλά νομίζω ότι αγωνιζόμαστε τώρα για τις ρυθμίσεις αυτές από τότε που άρχισα εγώ να είμαι ευρωβουλευτής και εγώ είμαι όσο το δυνατόν ένθερμος οπαδός τη μεταφορά από τον δρόμο στο σιδηρόδρομο. Εφόσον αυτό είναι δυνατόν, οφείλουμε να σημειώσουμε στην πολιτική μεταφορών ότι ούτε στην Κομισιόν, ούτε στο Συμβούλιο, αλλά ούτε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υπάρχουν πραγματικά πλειοψηφίες που να θέλουν όντως την μεταφορά από τον δρόμο στο σιδηρόδρομο. Και έτσι υπό τη σκοπιά αυτή έχουν επιτευχθεί πολλά πράγματα. Μακάρι να υπήρχαν και άλλοι πολιτικοί, όπως ο κ. Κράντες Πασχουάλ, ο οποίος λέει ότι όντω δεν το βρίσκει τόσο σκόπιμο, δεν το βρίσκει τόσο ευφυές και άλλα πράγματα γι' αυτόν είναι σημαντικότερα. Ας σταματήσουμε λοιπόν αυτή την υποκρισία να λέμε ότι θέλουμε μετακίνηση των μεταφορών από, το, τον δρόμο, τον αυτοκινητόδρομο, δηλαδή στο σιδηρόδρομο. Ας πούμε, δεν θέλουμε διότι δεν τη βρίσκουμε σκόπιμη τότε θα ήταν ειλικρινέστερη συζήτηση. Όμως όταν συζητούμε σήμερα για το ότι είναι απολύτως φυσιολογικό να πληρώνονται για τα τρία χρόνια πλήρως τα εξωτερικά στοιχεία κόστους και να, λέμε ότι είναι καλό το αποτέλεσμα εάν τα φορτηγά αυτοκίνητα πληρώνουν για παράδειγμα 10% ε, τότε κάτι δεν πάει καλά στη συζήτησή μας. Ίσως τότε πραγματικά να μην θέλουμε την μετακίνηση από το δρόμο στο σιδηρόδρομο. Όσοι είναι υπέρ αυτής της απόψεως, εγώ δεν είμαι, ας το πούν τουλάχιστον ευθαρσώς και ειλικρινά. Κυρία Μάισνερ, παρακαλώ δύο λεπτά. Είναι ο εφιάλτης του Προέδρου όταν ε, πλησιάζει το τέλος της συζητήσεως και όλο και περισσότεροι σηκώνουν τα χέρια. Θα προσπαθήσω να μην είμαι εφιάλτης για σας, για σας Πρόεδρε, λέει η κυρία Μάισνερ. Το κρίσιμο εν προκειμένου είναι ότι πραγματικά επιτέθηκαν πολύ λίγα. Ωστόσο ο κύριος Ελχαντράουι απέδειξε τις διπλωματικές του ικανότητες. Τουλάχιστον το καλό είναι ότι η θύρα παραμένει ανοιχτή για την ε, εσωτερήκευση των εξωτερικών ε, στοιχείων κόστους. Όλοι αγωνιστήκαμε υπέρ του earmarking για συγκεκριμένους σκοπούς Γι' αυτό εκφράζω τον σεβασμό για την προσπάθεια του ε, εισηγητού. Μπορεί να μην είναι πλήρες το αποτέλεσμα, αλλά τουλάχιστον είναι ένα βήμα. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, Πρόεδρε. Παρόλο που ζήτησα το λόγο κάπως αργά, ζήτησα το λόγο για να τονίσω το εξής. Το θέμα είναι άκρος ενδιαφέρον, το γνωρίζω αρκετά καλά. Άκουσα ε, για τους φιλόδοξους στόχους του τομέα, όμως τίνουμε να ξεχνάμε ότι μεταφορά αφορά εκατοντάδες χιλιάδες θέσεων εργασίας. Και τη στιγμή που θα υπάρχει επιπρόσθετο κόστος για τους ε, μεταφορείς, μπορεί να σημαίνει απολύσεις. Και αυτός το μέσο είναι στα όρια της κερδοφορίας, μην το ξεχνάμε. Επίσης αυτό, είπατε ότι τα οχήματα είναι παλαιά. Ναι, βεβαίως είναι παλαιά γιατί κανένας δεν μπορεί να αγοράσει ε, καινούρια. Οι εταιρείε αυτές ε, ε, αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες για να αντεπεξέλθουν. Δεν μπορούν να γίνουν νέες αγορές βαρέων οχημάτων. Μην ξεχνάμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε εκατοντάδες ε, χιλιάδες απολυμένους. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Και εν μία νυχτή μπορούν να απολεστούν αυτές οι θέσεις εργασίας. Βεβαίως όλοι λέμε ότι θέλουμε να ε, γίνουν επενδύσεις ε, σε νέα οχήματα και ούτω καθεξής. Ναι, οχήματα, σιγαστήρες και ούτω καθεξής, αλλά ε, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατήσουμε θέσεις εργασίας. Πρόκειται για ανθρώπους με πραγματικές ανάγκες. Πάλι καλά που ζήτησα τον λόγο μετά από την τελευταία αυτή παρέμβαση Υπάρχουν μελέτες που αποδείχνουν ότι στη Γερμανία ο φορολογούμενος πληρώνει επιδοτή κάθε θέση απασχόλησης στις οδικές μεταφορές με 3.000 ευρώ τον χρόνο και χωρίς να περιλαμβάνεται το κόστος για το περιβάλλον. Και τα 90% πληρώνει ο φορολογούμενος από τις ανάγκες αυτές. Γιατί διατηρούμε μια επιχείρηση, γιατί διατηρούμε με την έννοια αυτή τις μεταφορές αυτές με επιδοτήσεις παρόλο που είναι ο επιβλαβέστερος τρόπος μεταφοράς. Τώρα έρχομαι στην Πολωνία. Λέτε ότι στην Πολωνία λειτουργεί καλά η μεταφορά από τις οδικές ε, αρτηρίες. Από το 1990 η Πολωνία έχει κλείσει 25% των σιδηροδρομικών συνδέσεων. Έχει κλείσει τις έχει καταργήσει. Εκεί δεν υπήρξε απώλεια θέσεων απασχολήσεως. Ενώ θα μπορούσε να είχε φροντίσει για διατήρηση του περιβάλλοντος. Κουβέντα δεν λέτε για αυτά τα πράγματα. Μόλις πάει κανείς να θίξει τους αυτοκινητοδρόμους, δεν ξέρω εδώ τη Γερμανία, αλλά τουλάχιστον από το 1990 έχουμε κλείσει 17% του συνδρομικού δικτύου και όποιος θέλει να προστατεύει τις θέσεις απασχόλησης να μην βγάζει απ' έξω τις ε, οδικές μεταφορές. Κύριε Πασκερέλη, ας πάμε πίσω στην Ευρωβινιέτα. Τι έχει να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι έχει να προσθέσει. Λίγα, λίγα, πολύ λίγα, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαίρεται από το αποτέλεσμα, συγχαίρει και τον εισηγητή για το εξαίρετο έργο του. Το κείμενο είναι ισορροπημένο. Ήταν δύσκολο βέβαια να καταφέρουμε να συνδυάσουμε δύο διαφορετικές απόψεις. Έγινε όμως λίγο πολύ. Σίγουρα δεν είναι στο ύψος των προσδοκιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της αρχικής της πρότασης. Αλλά θέλω να το πω αυτό και σε όλους τους ευρωβουλευτές οι οποίοι εξέφρασαν επικρίσεις ότι δεν είναι αρκετά φιλόδοξο. Εγώ έχω να πω ότι το ποτήρι είναι κάτι παραπάνω από μισογεμάτο, γιατί υπάρχουν πολλές ε, γενικές αρχές που αναφέρονται εδώ μπορεί να υπάρξει εσωτερήκευση του εξωτερικού κόστους. Αυτό είναι πολύ βασικό και ευθυγραμμίζεται με την λευκή βίβλο που παρουσίασε η Επιτροπή πριν από μερικού μήνες. Αποτελεί τον μοχλό που θα επιτρέψει να εφαρμοστεί γενικότερα η αρχή αυτή σε όλες τις μορφές μεταφορών. Και το θέμα του earmarking τώρα. Είμαστε πιο φιλόδοξοι. Έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες από αυτά που είχαμε στο κείμενο του 6 υπάρχει ένα ολόκληρο άρθρο που αναφέρεται στους κανόνες για την εκχώρηση εσόδων. Ή γίνεται μια πρόταση για 15% τουλάχιστον των εσόδων που και από το εξωτερικό κόστος και από τα διόδια για τις υποδομές θα πηγαίνουν στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Και υπάρχει και υποχρέωση διαφάνειας για τα κράτη-μέλη χωρίς εδώ να παρεμβαίνουμε στο θέμα της φορολογικής κυριαρχίας των κρατών μελών, γιατί είδαμε ότι το Συμβούλιο δεν ήθελε να αλλάξει τίποτα. παρόλα αυτά υπάρχει δέσμευση από τα κράτη-μέλη ώστε να ενημερώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το κοινό και τα άλλα κράτη-μέλη για το τι γίνεται από τα έσοδα με τα έσοδα των διοδίων. Τα αντίστοιχα ποσά να είμαστε σίγουροι ότι πηγαίνουν στις μεταφορές. Έπειτα υπάρχουν και διάφορε τεχνικέ λεπτομέρειε, ανέφερε και ο συγγετή. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να ετοιμάσει ένα εγχειρίδιο, έναν οδηγό για τι διακυμάνσει των ε, ε, τελών, είτε λόγω συμφόρεση είτε υποδομών. Υπάρχει ένα πακέτο που ενθαρρύνει επίσης την ανανέωση των οχημάτων αναφέρονται επίσης και εξαιρέσεις για τα νέα οχήματα, αλλά αναφέρονται επίσης και κυρώσεις για τα οχήματα που ρηπαίνουν περισσότερο. Υπάρχει μια πραγματική υποχρέωση προσδιορισμού με διατάξεις του ΜΑΚΑΠ Και υπενθυμίζω εδώ επίσης ότι πρόκειται για τη δουλειά που θυμίζει τον ιστό που ήφαινε η Πινελόπη. Από το 2006 έχουμε ξεκινήσει, το 2008 προχωρήσαμε, το 2011 είχαμε μια πρώτη έκθεση, υπάρχει και επόμενη της Κομισιόν του χρόνου. Σε τέσσερα χρόνια περιμένουμε νομοθετική πρόταση. Είναι δηλαδή ένας τομέας στον οποίο προχωράμε σιγά σιγά γιατί πολιτικά είναι πολύ ευαίσθητα τα ζητήματα που συζητάμε. Συνεχίζουμε πάντως να προδεύουμε. Πρέπει να δούμε τι πρόοδο έχουμε πετύχει μέχρι τώρα και να μην κοιτάμε μόνο το επεισόδιο Ευρωβινιέτα. Ελπίζω η ψηφοφορία του Κοινοβουλίου στις 8 Ιουνίου να είναι υπέρ του κειμένου αυτού. Γιατί τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανοίγει το δρόμο σε μια πραγματική εσωτερήκευση του εξωτερικού κόστους για τις μεταφορές και όχι μόνο. είναι η μαρτυρία μιας πραγματικά βιώσιμης πολιτικής μεταφορών που διασφαλίζει την κινητικότητα, φροντίζει για την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ε, τώρα δεν ξέρω να συμμερίζουμε την άποψή σας ότι το ποτήρι είναι κάτι περισσότερο από γεμάτο. Εγώ θα έλεγα απλώ ότι δεν είναι άδειο. Αλλά έχει περισσότερο ε, νόπνευμα παρά ουσία το 1% του κάτι είναι προτιμότερο από το 100% του τίποτα. Και με αυτό είχαμε να κάνουμε μέχρι τώρα. Κύριε Σιγητά, πολύ σύντομα θέλετε να πείτε κάτω γιατί μας περιμένει και ο κύριος Ρόιτερ για τα ποτά. Δύο λεπτά παρακαλώ. Τίποτα παραπάνω. Μπορεί και λιγότερο. Ένα λεπτό. Ναι. Το μόνο που ήθελα εγώ να πω είναι ευχαριστώ τους συναδέρφους για τα σχόλιά τους, για τη στήριξή τους. Με τη στήριξη αυτή μπορέσαμε να προχωρήσουμε και να κάνουμε το Συμβούλιο να μετακινηθεί. και να πετύχουμε έστω και με μικρή πλειοψηφία από το Συμβούλιο το Συμβασμό αυτών. Για το earmarking. Η Κομισιόν λέει ότι είναι κάτι παραπάνω από αυτό που νομίζουμε. 15% λέει η συμφωνία των εσόδων πρέπει να πηγαίνει στα διευρωπαϊκά δίκτυα και στις μεταφορές. Είναι παραπάνω από το σύνολο του εξωτερικού κόστους. Αν τα βάλετε και τα δύο μαζί, είναι πολύ. Δηλαδή εμείς μπορούμε να πούμε ότι όλα τα έσοδα από το εξωτερικό κόστος τελικά θα πηγαίνουν στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Σε σχέση με το τι είχαμε μέχρι τώρα, όπου δεν είχε προβλεφθεί τίποτα γι' αυτό, είναι μια μεγάλη πρόοδος. Έπειτα υπάρχει και το θέμα τη διαφάνεια, που είναι υποχρεωτική ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να το αποδεικνύουν ότι τα έχουν δώσει αυτά τα λεφτά στι μεταφορέ. Τέλο, είναι ένα σημαντικό βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Δεν είναι το τέλο τη διαδικασία, όχι. Αλλά μέσα στο πλαίσιο το πολιτικό στο οποίο λειτουργήσαμε, πιστεύω ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ πολύ όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή και τους και εισηγητές για την δουλειά καθώς και το προσωπικό και της γραμματείας. Πρόκειται για το τελευταίο θέμα που χειρίστηκε η Βανέσα. Όχι στο Κοινοβούλιο βέβαια, αλλά για, την, για λογαριασμό της Επιτροπής Μεταφορών. Και θα πάνε στην Επιτροπή σε άλλη επιτροπή, σε άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή και η ψηφοφορία θα γίνει στις 7 Ιουνίου, Τρίτη. Δύσκολο και το θέμα, δύσκολες και διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι και τον εισηγητή και, τις, και τους κοιόδες εισηγητές. Ακολουθεί τώρα η ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών, ανταλλαγή με, απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ας έρθει ο κύριος Ρόιτερ εδώ για να τον έχουμε πιο κοντά μας ως πλέον εύκολο στόχο για μια συζήτηση που υπόσχεται να είναι πολύ ζωηρή. Καλά λοιπόν, κύριε Ρόιτε, τι θα μας πείτε. Παρακαλώ εσείς, συνάδελφοι, ήρεμοι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα είναι χαρά μου να είμαι εδώ κοντά σας, ιδίως μετά από το έσιον πέρας των διαπραγματεύσεων για την Ευρωβινιέτα. Βέβαια το δικό μου θέμα είναι πιο δύσκολο. Θα σας ενημερώσω σχετικά με το πού βρισκόμαστε για το θέμα των υγρών. Α, ναι, ναι. Σηκώνει την κάρτα του ο ε, Ευρωβουλευτής για να σημειωθεί το όνομά του να μπορέσει μετά να παρέμβει. Θα σας πω λοιπόν για το θέμα των υγρών. Είχα ήδη την ευκαιρία και νομίζω οι περισσότεροι εξημών γνωρίζετε. Έχω συζητήσει δύο φορές ήδη με τους συντονιστές στις 3 και στις 10 Μαΐου Εν τέλει πάντως είχαμε πει να έλθει εδώ, να έλθω εγώ εδώ ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μιλήσω σε ολόκληρη την Επιτροπή. Πρώτα πρώτα ζητεί συγγνώμη ο κύριος Κάλλας, το συζήτησα χθε το θέμα μαζί του, πολύ θα ήθελε να είναι παρόν, αλλά για την ώρα κάνει μια δουλειά που θα εκτιμήσετε και εσείς. Συζητεί δηλαδή με τους υπόλοιπους επιτρόπους την επόμενη δημοσιονομική πολυ, ετή δημοσιονομική προοπτική, άρα κολλείεται και με παρακάλεσε να εμφανιστώ εγώ εδώ ε, ε, εκπροσωπώντας τον. Πού βρισκόμαστε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία ημέρα πριν από τις 29 Απριλίου υπέβαλε σύσταση προς τις χώρες μέλη να αναβάλουν την εισαγωγή της χαλάρωσης των ελέγχων των υγρών ε, duty free που έχουν αγοραστεί σε τρίτες χώρες μέσα σε ε, ασφαλισμένες σακούλες. Γιατί αυτό? Διότι ήταν σαφές, πολύ σαφές, τις τελευταίες δύο εβδομάδες πριν από το τέλος Απριλίου, ότι μεγάλος αριθμός χωρών μελών δεν θα εφάρμοζαν το θέμα αυτό Ε, είχαμε φτάσει σε έναν αριθμό μεγαλύτερο από το μισό των χωρών μελών. Μια ε, πραγματικά πολύ ανησυχητική κατάσταση. Είχαμε συζητήσει, αν θυμάστε, σχετικά με το ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να παραμείνει, να εμείνει στις θέσεις της για την εισαγωγή χαράρωσης των ελέγχων υγρών, διότι θεωρούσαμε ότι λίγες μονοχώρες θα αντιτίθετο. Εν τέλει ωστόσο είχαμε απέναντί μας 15 περίπου χώρες μέλη και ταυτόχρονα μία ημέρα πριν από την υποτιθέμενη εισαγωγή της ρύθμισης αυτής έτοιμα να γίνει διαβούλευση για τους ελέγχους ασφαλείας για τα υγρά τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες. Έτσι λοιπόν, εξ ονόματος του κυρίου Κάλλας ήρθα σε επαφή με τον πρόεδρό σας που είπε ότι για λίγες ημέρες ή λίγες εβδομάδες θα μπορούσαμε ίσως να δεχθούμε αναβολή της εφαρμογής του μέτρου, αλλά μόνο για λίγες εβδομάδες και εμείς έκτοτε ε, είμαστε στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσουμε. Πού βρισκόμαστε τώρα. Πρώτα, μετά από την κοινοποίηση από τις Ενωμένε Πολιτείες ζητήσαμε αμέσως ε, να έλθει διαπραγματευτής από τις Ηνωμένε Πολιτείες στις Βρυξέλλες να μας μιλήσει για τα πρόσθετα μέτρα ελέγχου τα οποία θα απαιτούσαν οι Ηνωμένε Πολιτείες όταν θα ε, προχωρούσαμε εμείς στην χαλάρωση των μέτρων αυτών. Αυτό το κάναμε στις 4 Μαΐου. Δυστυχώς οι συζητήσεις που διεξαγάγαμε οδήγησαν στο ότι στις 6 Μαΐου η συμφωνία όπου είχαμε καταλήξει καταρχήν με τον διαπραγματευτή δεν έγινε αποδεκτή για λόγους ασφαλείας όπως μας είπε η Ουάσιγκτον και ιδίως ε, λόγω των, ε, της καταστάσεως ασφαλείας μετά τον θάνατο του Μπιν Λάντεν και έτσι στις 12 Μαΐου συζητήσαμε την κατάσταση με τις χώρες μέλη από τις εννέα χώρες μέλη που ήταν έτοιμες και διατεθειμένες να προχωρήσουν στην χαλάρωση των μέτρων ελέγχου των υγρών πρώτον, πρώτου τέλους Απριλίου μόνο δύο έως τρεις εξακολουθούσαν να είναι διατεθειμένες εάν αυτό σημαίνει να υποχρεώσει να λαμβάνουν ε, αυστηρά μέτρα ελέγχου για υπερατλαντικές πτήσεις. Βρισκόμαστε τώρα στην δύσκολη ομολογουμένως κατάσταση να έχουμε 25, 24, 26, 24 έστω χώρες μέλη οι οποίες πιθανόν θα χρησιμοποιήσουν αυτή την let out clause που λέτε εσείς δηλαδή ρήτρα που προβλέπει νομοθεσία και που επιτρέπει σε κάθε χώρα μέλος να εφαρμόζει αυστηρότερα μέτρα. Βέβαια, θα μπορούσαμε να κάνουμε το τεστ, να δούμε αν όντω είναι πιο αυστηρά τα μέτρα με 24 χώρες μέλη. Αλλά καταρχήν και δοθήσεις της καταστάσεως ασφαλείας που αντιμετωπίζουμε σήμερα θα ήταν δύσκολο το εγχείρημα αυτό. Άρα εσωτερικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον Αντιπρόεδρο Κάλλας καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι πιθανώς χρειάζεται να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από μια δύσκολη κατάσταση, να χρησιμοποιήσουμε την κατάσταση αυτή έτσι ώστε να προετοιμάσουμε καλύτερα την προσπάθεια επίτευξης του πραγματικού μεγάλου στόχου της κατάργησης δηλαδή των ελέγχων των υγρών για την οποία στοχεύουμε μέχρι το 2013. Αυτό λοιπόν που θα θέλαμε να προτείνουμε τώρα, να σας προτείνουμε, είναι να προχωρήσουμε σε μια προσπάθεια αλλαγής των υφισταμένων κανόνων και μετατροπής μιας υποχρέωσης να εισαχθεί μια χαλάρωση των μέτρων ελέγχου για τα εισαγόμενα υγρά από τρίτες χώρες να το τροποποιήσουμε ώστε να γίνει ένα δικαίωμα, όχι πλέον υποχρέωση, αλλά δικαίωμα για τις χώρες μέλη να το πράξουν, άρα να έχουν την επιλογή οι χώρες μέλη αν θέλουν να το πράξουν ή όχι. Δεν είναι υποχρεωμένες να λάβουν αυστηρότερα μέτρα για να μπορέσουν να κάνουν αυτό το opt-out, Όσε όμως θεωρούν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν πιο χαλαρά, να εφαρμόσουν πιο χαλαρά μέτρα, όσες δεν έχουν υπερατλαντικές πτήσεις, όσε έχουν άλλο εξοπλισμό και θέλουν να ε, ελέγξουν την δράση του, να κάνουν τεστ δηλαδή, αλλά η ολοκληρωτική κατάργηση των ελέγχων για τα υγρά να παραμείνει ο απότερος στόχος του 2013. Εσείς θα μου πείτε τώρα, ε, μάλλον θα με ρωτήσετε τι μας διασφαλίζει ότι δεν θα βρεθούμε στην ίδια κατάσταση του 2013 όπως βρισκόμαστε τώρα. Το μόνο που μπορώ να πω εν προκειμένου είναι ότι διδαχθήκαμε από τις πρόσφατες εμπειρίες μας και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι αντί να εμπιστευόμαστε, καλύτερα να ελέγχουμε. Άρα να προτείνουμε καταρχήν να κινηθούμε προς την κατεύθυνση της προθεσμίας 2013, να ορίσουμε γρήγορα μια ομάδα εργασίας με συμμετοχή χωρών μελών, με συμμετοχή εκπροσώπων του κλάδου που ε, κατασκευάζει τα σχετικά μηχανήματα για τον ελέγχο των υγρών με τα αεροδρόμια, με τις αεροπορικές εταιρείες, αλλά βεβαίως και με εσά και δίνοντάς σας το λεγόμενο feedback σε μόνιμη βάση για το ποια μορφή θα λάβει αυτός ο οδικός χάρτης μέχρι την τελική κατάργηση των ελέγχων του 2013 ώστε να μην φτάσουμε λίγες εβδομάδες ή μόνο λίγες ημέρες πριν από την εφαρμογή της χαλάρωσης όπως έγινε την προηγούμενη φορά όπου είχαμε την εντύπωση ότι ίσως λίγες χώρες να καθυστερούν πάλι λοιπόν να μην βρεθούμε εκτός πραγματικότητας άρα ίδρυση ομάδας εργασίας ενημέρωσή σας διαρκής ενημέρωση με τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι το 2013 θα είναι η σωστή προθεσμία. Επίσης, να μην μας έρθει καμία έκπληξη από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Θα θέσουμε το θέμα λοιπόν και στα πλαίσια της Επιτροπής Ανοιχτών Ουρανών, Open Skies Committee, που θα συνέλθει στις 23 Έκτου και να κινηθούμε προς την κατεύθυνση μιας κοινής Δήλωση Ενωμένων Πολιτειών Ενωμένης Ευρώπης για μια συνεργασία για ολοκληρωτική κατάργηση των ελέγχων των υγρών μέχρι το 2013. Το 2013 μάλλον. Είμαι βέβαιος ότι όλα αυτά είναι σημαντικά. Ασφαλώς μπορείτε να με επικρίνετε, να μου πείτε ότι θα έπρεπε να τα είχα σκεφτεί αυτά το 2011. Νομίζω ότι δεν έχει βέβαια νόημα τώρα να ακυρώσουμε την προθεσμία του 2013, αλλά πρέπει να την επανεξετάσουμε με ξεκάθαρο και επίμονο τρόπο ε, τους επόμενους μήνες, ίσως και το 2012, και να δούμε αν όντως έχει, είναι σκόπιμη. Αλλά νομίζω ότι αυτό θα λέγαμε ότι είναι το καλύτερο να κάνουμε. Βεβαίω και δεν υπερηφανεύομαι για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, είμαι και εγώ αλλά και ασφαλώς ο Αντιπρόεδρος ε, κύριος Κάλλας ιδιαίτερα αναστατωμένοι από την πορεία αυτή ότι δεν μας είχαν ενημερώσει οι χώρες μέλη, δεν είχαμε προειδοποιηθεί επαρκώς και εγκαίρως με σωστό τρόπο από τους υπερατλαντικούς εταίρους μας, οι δε μηχανισμοί που θα θεσπίσουμε τώρα θα πρέπει να είναι τέτοιοι που να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρχει και η ενημέρωση αλλά και ο έλεγχος αυτός. Αυτά μπορώ να πω κύριε Πρόεδρε και είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν πολλές ερωτήσεις. Θα δώσω στα μέλη τρία λεπτά στον καθέναν έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα... Ε, De Grandes Pascal, Mr. Leakfried, Mr. Zasada and Mr. Fleckenstein. Is that it? Έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να απαντήσουμε. Και εγώ στο τέλος θα μιλήσω για να βάλω το κερασάκι στην τούρτα. Γκρός. Είχαμε ήδη την ευκαιρία να συζητήσουμε. Βεβαίως εγώ θα προτιμούσα αντί της Κομισιόν να βρίσκεται ενώπιον μας το Συμβούλιο. Εκεί χρειάζεται να διευκρινιστούν ορισμένα πράγματα για το μέλλον. Εν μέρη συμφωνώ με την ανάλυση σας, αν και γνωρίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε αξιώσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν ήδη η Γαλλία είχε ανακοινώσει ότι αντιμετώπιζε προβλήματα, είχαμε θέσει το ερώτημα τι θα γίνει εάν και οι άλλε χώρε αντιδράσουν με τον ίδιο τρόπο. Και είτε το θέλουμε είτε όχι, μπαίνουμε σε μια κατάσταση η οποία δημιουργεί ένα προηγούμενο. Και αυτό το προηγούμενο σημαίνει πολύ απλά ότι το Συμβούλιο δεν πληρεί τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Και βέβαια ανοίξαμε και ένα παράθυρο για να προσδώσουμε νομότυπο χαρακτήρα σε μια παρανομία. Και είπατε κι εσείς ότι πρέπει να τονίσουμε στο Συμβούλιο κανείς εξημών δεν θεωρεί ότι είναι θέμα ασφαλείας. Είναι θέμα του ότι οι χώρες δεν θέλουν να επενδύσουν. Και ξαναρχόμαστε στην ίδια παλαιά συζήτηση. Όταν πρόκειται για θέμα ασφάλειας των αεροδρομίων, ποιος είναι αυτός που πληρώνει. Και αυτό είναι το θέμα γύρω από το οποίο στρέφεται η συζήτηση. Δεύτερο, η συζήτηση αυτή δεν είναι ανέντιμη μόνο απέναντι στο κοινοβούλιο, είναι ανέντιμη απέναντι και στους επιβάτες, διότι μειώνει το επίπεδο ασφάλειάς τους. Και τέλος είναι ανέντιμη και απέναντι στα αεροδρόμια, τα οποία ήδη έχουν προβεί σε επενδύσεις. Και η απόφαση που λαμβάνεται τώρα δεν ανταποκρίνεται σε αυτές, στις προσδοκίες αυτών των τριών φορέων που ανέφερα. Ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα βεβαίως και εμείς επιθυμούμε να συνεργαστούμε ώστε να υπάρξει μια θετική έκβαση. Ωστόσο, συνάγουμε συμπεράσματα. Δεν θέλουμε πλέον ρήτρα opt-out για αποφάσεις οι οποίες έχουν σχέση με ασφάλεια. Γιατί η κατάχρησή της θα γίνει οπωσδήποτε στο μέλλον. Δεύτερο, πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε διασύνδεση με την τεχνολογία. Έχουμε δει και στο παρελθόν ότι βάζουμε προθεσμίες ελπίζοντας ότι θα προκύψει η απαραίτητη τεχνολογική λύση και μετά αναθεωρούμε τις προθεσμίες αυτές διότι δεν έχει ακολουθήσει η τεχνολογία. Τρίτο, σε ό,τι αφορά συμφωνίες με τρίτες χώρες, εν προκειμένου Ηνωμένε Πολιτείε θα πρέπει να δεσμεύονται αυτές εκ των προτέρων. Εγώ δεν έχω πρόβλημα τώρα να θεωρήσουμε το έτος 2011 ως επιλογή. Εγώ θα προτιμούσα το 2012 ανεξαρτήτως αποφάσεως για το 2013 να έχουμε τη δυνατότητα, να έχουμε την ευκαιρία να συνεννοηθούμε με όλους τους ενδιαφερομένους εταίρους και επομένως και με τις Ενωμένες Πολιτείες για να λάβουμε απόφαση για το πώς θα προχωρήσουμε πλέον το 2013. Δεν θέλω να ληφθεί σήμερα απόφαση για το 2013, διότι κατόπιν θα αμφισβητηθεί είτε για λόγους τεχνολογικούς, είτε για λόγους ασφαλείας, είτε με τα ίδια επιχειρήματα με τα οποία αμφισβητήθηκε το 2011. Αν θέλουμε λοιπόν να διατηρήσουμε κάποια αξιοπιστία εδώ της Ευρωβουλής, θέλω και το 2012 να υπάρξει μια ημερομηνία όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα λάβουν αποφάσεις το 2013. Ερχαντράουι, τρία λεπτά. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Είμαι συντονιστή, οπότε είχα την ευκαιρία να συζητήσω και για κλεισμένο το θυρών μαζί σας. Είναι η δεύτερη φορά πάντως που αναβάλλεται η υπόθεση αυτή. Και υπάρχει κριτική πάντα που λέει ότι την τελευταία στιγμή δεν θέτουμε σε εφαρμογή το μέτρο. Η Επιτροπή είχε πρόβλημα μεθοδολογίας και η ιδέα της ομάδας εργασίας δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί μέχρι τώρα. Εν πάση περιπτώσει, ας κοιτάμε τώρα προς τα μπρος και ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει κατάχρηση για την εφαρμογή αυτή από τα κράτη-μέλη ώστε να εφαρμόσουν ακόμα πιο αυστηρά μέτρα. Πρέπει να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα προς τα κράτη-μέλη και σε σχέση με την έκθεση Lightfrit που έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση των πιο αυστηρών μέτρων, ότι θα έχουμε δέσμευση από το Συμβούλιο ότι θα πάρει στα σοβαρά αυτή την υπόθεση και ότι θα καταλήξει κάπου. Δεν θα τον μπλοκάρει συνέχεια. Επιτέλους, ήρθε η στιγμή να στείλουμε αυτό το ισχυρό μήνυμα. Κατά τα άλλα, ναι, δεδομένη της λιβερής κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε, πιστεύω ότι κάτι είναι και αυτό. Ας επικεντρωθούμε στην ημερομηνία του 2013. Η πρόταση που κάνετε, ε, να βάλουμε και τους Αμερικανούς μέσα, ναι, πολύ καλό, ναι, αλλά θα ήθελα και δέσμευση από το Συμβούλιο. Να έχουμε ίσως μια ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα έξω που να συμπεριλαμβάνει και την Προεδρία, ώστε ανοιχτά να δεσμευθεί και το Συμβούλιο για την ημερομηνία του 2013. Ελπίζουμε να δουλέψουμε και εμείς μαζί με την ομάδα αυτή εργασίας, επιμονή μου βάσεως, ώστε να παρακολουθήσουμε από κοντά την υπόθεση αυτή και όχι μόνο μερικές εβδομάδες πριν τη λήξη της προθεσμίας ε, ξαφνικά να μπαίνουμε στο παιχνίδι και να βλέπουμε τα προβλήματα. Η Μάισνερ. Ευχαριστώ. Αρνούνται οι χώρες μέλη. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάτι έχει εγκριθεί και μετά δεν προχωρεί. Φαίνεται παράλογο γιατί εδώ μιλούμε εν πάση περιπτώσει για την διευκόλυνση της ζωής των πολιτών. ελαφρύνσης δηλαδή. Είναι κρίμα που δεν έγινε αυτό που ότι θα γινόταν στις 29 Απριλίου. Βεβαίω μόνο οι insider τα γνωρίζουν αυτά, δεν τα γνωρίζουν όλοι. Οι επιβάτες δεν τα γνωρίζουν αυτά πράγματα, οπότε δεν υπάρχει και μεγαλύτερη ζημιά αξιοπιστίας. Η ζημιά περιορίζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια, δημιουργείται και προηγούμενο, όπως είπε ο Ματιό Για μένα το ερώτημα είναι εάν ο κλάδος, η βιομηχανία δηλαδή, η οποία κατασκευάζει τα μηχανήματα αυτά, εάν θα πρέπει να συμμετάσχει σε αυτή την ομάδα εργασίας ή αν απλώς θα πρέπει να προσκαλείται να εξηγεί που βρίσκεται τεχνολογικά. Οι συζητήσεις με τις ΗΠΑ μου φαίνονται σωστές, μου φαίνεται σωστό δηλαδή να, γίνει ε, αυτό και προσπαθώ να δω θετικά τα πράγματα. Ίσως είναι θετικό για το 2013 όπου πραγματικά η τεχνολογία θα είναι κατά πολύ βελτιωμένη, η τεχνολογία που θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ώστε να διευκολυθούν πολύ οι ε, έρευνες, η έλεγχοι. Οι διάφοροι σαρωτές θα έχουν βελτιωθεί και ίσως τελικά η λύση να είναι λογική. Λίχτενμπεργκερ, τρία λεπτά. Θα συμφωνήσω σε πολλά με τον ε, συνάδελφό μου, κύριο Γκρός. Το πρόβλημα είναι απλό. Όταν θα υπάρχει ρήτρα opt-out, θα χρησιμοποιηθεί. Αυτή τη φορά μάλιστα με υπερβολικό τρόπο. Αλλά όλο και περισσότερο το Συμβούλιο δεν ενδιαφέρεται πλέον να έχει ευρωπαϊκές ρυθμίσεις. Προτιμούν οι περισσότεροι να παίζουν το παιχνίδι μόνοι τους και οι υπόλοιποι προτιμούν να αρπάξουν τα λεφτά και να το βάλουν στα πόδια, με λίγα λόγια. Αυτό να μην το λησμονούμε και για, το όσα θα, για τα όσα θα πράξουμε στο μέλλον και για τον σχεδιασμό, για το πώς θα προχωρήσουμε πραγματικά το 2013. Συμφωνώ με την φίλη μου κυρία Μάισνερ και γι' αυτό λέω ότι αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία θα διαπραγματευτεί η βιομηχανία με την Κομισιόν, αλλά αυτοί οι οποίοι πληρώνουν, αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνουν το κόστος και θα συζητήσουν με τους ειδικού της ασφάλειας, με τους ειδικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι έχω βαρεθεί πλέον να μας υπαγορεύουν άλλοι το ποια μηχανήματα θα χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον. Ναι, υπάρχουν συσκευές οι οποίες μπορούν να ανακαλύψουν σχεδόν τα πάντα, είναι όμως και υπερβολικά δαπανηρές. Όποιος ισχυρίζεται ότι μπορεί να ανακαλύψει τα πάντα, σε έναν έλεγχο δηλαδή, θα πρέπει να εξηγήσει και πόσο θα κοστίσει αυτό. Βεβαίω και υπάρχουν τεχνολογίε. Αλλά πρέπει να είναι σαφέ ότι υπάρχει και υψηλό κόστο. Εγώ νομίζω ότι η δυνατότητα αυτή που περιγράψατε είναι και η μοναδική, διπυρό μεν, αλλά έτσι είναι, η πορεία αυτή δηλαδή. Νομίζω ότι για το 2012 θα χρειαστούμε μια ξεκάθαρη αξιολόγηση και σε ό,τι αφορά την αναγκαιότητα των κανόνων ασφαλείας αυτών. Και το έχουμε συζητήσει και την τελευταία φορά, από την άποψη δηλαδή της χημίας. Τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα. Αυτή την αξιολόγηση, αυτό το assessment θέλω να το δω πρώτα. Και μετά να συζητήσουμε με βιομηχανία, με κατασκευαστές και ούτω καθεξής. Θέλω να δω, πραγματικά πρόκειται για την απειλή νούμερο 1, την πιο σημαντική απειλή Βεβαίω και πρόκειται και για θέμα κόστου. Και το ερώτημα του κόστου πρέπει να το συζητήσουμε. Διότι αλλιώ θα πέφτουμε διαρκώ στην ίδια παγίδα. Για ένα θέμα θέλω να λάβω θέση ακόμη. Θα γίνει συνάντηση τη Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκή Ένωση με Ηνωμένε Πολιτείε στην Βουδαπέστη. Όπου κατά πάσα πιθανότητα θα συζητηθεί όχι μόνο το PNR αλλά και όλα τα θέματα ασφαλείας δηλαδή η διαβίβαση των ε, προσωπικών δεδομένων των επιβατών, αλλά και όλα τα άλλα θέματα ασφαλείας της αεροπορικής μεταφορές. Ας ξεχάσουμε την προσπάθεια να μεταφέρουμε με το λεγόμενο copy-paste ό,τι ρύθμιση έχουν λάβει οι ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας δείξουμε κάπως μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, διότι αλλιώ θα βρισκόμαστε ξανά και ξανά στην ίδια κατάσταση. Κάτι το οποίο βεβαίως δεν ε, είναι καλό για την ευρωπαϊκή αξιοπιστία. Φώστερ, τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις επεξήσεις από τον κύριο Ρόιτερ. Θα ήθελα να πω ότι δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε από εμά θα πίστευε ότι θα μπορούσαμε μέχρι τις 29 Απριλίου 11 να δεχτούμε αυτό το πλαίσιο. Μιλήσαμε με τους κατασκευαστές, ξέρουμε κατά πόσο μπορούν να ανταποκριθούν. Θα ήταν πολύ θετικό, αλλά νομίζω ότι το 2013 είναι πιο ρεαλιστικό. Προσωπικά πιστεύω ότι θα ήταν άκρος αφελές να θεωρήσετε ότι όλα τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να συμμορφωθούν, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι τα διάφορα κράτη-μέλη έχουν διάφορα επίπεδα αντιμετώπισης απειλών, κάτι το οποίο δεν θα αλλάξει. Γι' αυτό, ως προς το θέμα μας, όταν ε, έγινε λόγος για το 2011 θα ήταν άκρος θετικό, αλλά εγώ επιβάτες και όλοι οι άλλοι δεν θα πρέπει να στέκομαι για τρεις-τέσσερις ώρες στο, ε, στην ουρά για να περάσω τη, στην ασφάλεια επειδή κάποιος ε, θεωρεί ότι μπορεί να προβάλλει νέα τεχνολογικά μέσα όλοι μπορούμε να δεχτούμε τα 100 μιλιλίτρ. Επί του παρόντος, μέχρι ότου είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει κατάλληλη τεχνολογία, όλοι έχουν την ε, κατάλληλη εκπαίδευση και μπορεί κάθε αεροδρόμιο να είναι λειτουργικό. Μπορείτε να μιλήσετε με τους Αμερικανούς. Μπορούμε να έχουμε μία ομάδα εργασίας. Θα πρέπει ο τομέας της βιομηχανίας να συμμετάσχει οι κατασκευαστές, τα αεροδρόμια, οι αεροπορικές εταιρείες, γιατί αν εγώ επιβιβαστώ στο αεροπλάνο θέλω να είμαι σίγουρη ότι είμαι ασφαλής σε 37.000 στα 37.000 πόδια. Γι' αυτό ας κάνουμε ένα βήμα προς τα πίσω για να προχωρήσουμε επικοδομητικά πιστεύω ότι μιλάτε με τους σωστούς ανθρώπους και θα ήταν σκόπιμο να προωθήσετε αυτές τις ζητήσεις και στο μέλλον να μας δώσετε πληροφορίες για να δούμε πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε λογικά. Ο κύριος Ντεγκράντες, για τρία λεπτά. Χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο κύριος ε, Ρώσα όρισε την ε, θέση της ομάδας μας και δεν θα αντιταχθώ σε αυτήν. Σύμφωνο απόλυτα. Θα ήθελα να εκφράσω μία σύντομη σκέψη. Διότι ήμουν εισηγητής της έκθεσης για την αεροπορική ασφάλεια. Σήμερα σε μια συνέντευξη τύπου έγινε λόγος για το γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε το, την προθεσμία της 29ης Απριλίου 2011. Ειλικρινά κύριε Ντερόιτερ, καταλαβαίνω ότι περνάτε μία δύσκολη στιγμή και δεν φέρετε καμία ευθύνη σε αυτή την ικτρή, κατάσταση. Αυτό με ενδιαφέρει είναι το γόητρο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Πρόκειται για μια παλαιά ιστορία. Καταρχήν εγκρίναμε ένα ψήφισμα το οποίο δεν υπερψήφισα εγώ που μιλήσαμε για, την, για το ότι καταδικάσουμε την τρομοκρατία γενικότερα. Και στη συνέχεια ζήσαμε μια άλλη ιστορία, φτάσαμε σε συμφωνίες και δεν μπορέσαμε να αρκεστούμε στα δεδομένα του παρελθόντος. Χρειάστηκε να κάνουμε, σε ένα, να κάνουμε ένα συμβασμό. Δεν πρέπει οι πολίτες να θεωρήσουν ότι η Κομισιόν, το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη ακολουθούν διαφορετικές όδους, διότι υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα και δεν υπάρχουν κοινές ευθύνες σε θέματα ασφάλειας. Δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτή η αντίληψη. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Εγώ βεβαίως θαυμάζω τι είπα, αλλά θα ήθελα να πω ότι όταν λαμβάνουν αποφάσεις δεν μας ρωτούν, τις λαμβάνουν και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τους ακολουθήσουμε. Σε αυτή την περίπτωση, εάν έχουμε μία ενιαία απόφαση, ελπίζω να είμαστε στο ύψος των περιστάσεων και να ε, σεβαστούν την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως θα έπρεπε. Πρέπει να λαμβάνουμε κοινέ αποφάσεις, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γόητρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ε, έγινε και τίποτα αυτό είναι ένα συμβάν, αλλά θα πρέπει τα, τρία θεσμικά όργανα να είναι στο ύψος των περιστάσεων, διότι οι πολίτες μας παρακολουθούν και απαιτούν από μας υπεύθυνε αποφάσεις. Η ασφάλεια αφορά θέμα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εμείς ε, λαμβάνουμε σοβαρές αποφάσεις υπέρ του Ευρωπαίου πολίτη και υπέρ της ασφάλειας. Ας είμαστε στο ύψος των περιστάσεων, διότι κάτι τέτοιο επιβάλλεται. Λάχτφριντ, για τρία λεπτά όλοι σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν μου αρέσει να αντίπω σε ορισμένους συναδέλφους και εν προκειμένου στην κυρία και δεν το πράττω καθόλου Ευχαρίστω. Δεν θεωρώ όμω ότι φταίει μονάχα το Συμβούλιο. Όλων η απόδοση έχει, είναι ελληματική. Όλων η προσπάθεια είναι ελληματική. Και των χωρών μελών αλλά ούτε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέδωσαν όπως έπρεπε. Εγώ είχα συμφωνήσει τότε με την ενδιάμεση λύση, αναλαμβάνω τις ευθύνες μου, αλλά δεν ήταν καλή ιδέα. Θεωρώ επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διάβασε σωστά τα σημάδια, εάν τα είδε. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μόλις μία ημέρα πριν από την υποτιθέμενη έναρξη της νέας φάσης δεν γνώριζε ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Μιλώ για τη χώρα μου, την Αυστρία. Δεν είχαν κουνήσει ούτε το μικρό τους δαχτυλάκι οι Αυστριακοί για να προμηθευτούν μηχανήματα, συσκευές και ούτω καθεξής. Ίσως θα έπρεπε να είχαμε αντιδράσει όλοι νωρίτερα. Ωστόσο θα συμφωνήσω εδώ με την κυρία Φώστερ θα πρέπει να καθίσουμε να συγκεντρώσουμε την προσπάθειά μας να δούμε ποια πράγματα είναι εφικτά και στη συνεργασία με τις χώρες μέλη αλλά και με τους υπερατλαντικούς εταίρους μας οι οποίοι θα, θα συμμετάσχουν με κάποια μορφή. Το χειρότερο νομίζω είναι να ξαναβάλουμε μια καθορισμένη ημερομηνία και πάλι δύο μέρες πριν από την ημερομηνία αυτή να βρούμε ότι πάλι δεν λειτουργεί. Το σύστημα που ισχύει τώρα λειτουργεί. Εάν εν πάση περιπτώσει ορισμένα καταστήματα αφορολογήτων κερδίζουν λιγότερα τώρα, ε, τι να κάνουν, μας κερδίσουν λιγότερα. Θα πρέπει να αντικαταστεί το σύστημα αυτό μόνο από ένα άλλο σύστημα που θα γνωρίζουμε ότι λειτουργεί, ότι τα μηχανήματα λειτουργούν και ούτω καθεξής. Αλλιώς δεν έχει, δεν έχει νόημα να αντικαταστήσουμε το σύστημα με ένα άλλο που δεν θα λειτουργεί. Ας δούμε λοιπόν ποιες ή θα είναι οι εξελίξεις, ας μην δεσμευτούμε με προθεσμίες που πάλι θα μπορέσουμε να τηρήσουμε, διότι πλέον κανείς δεν θα μας παίρνει στα σοβαρά. Ο κύριος Σάντα, τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμφωνώ με τον κύριο Λάκτριτ, τον προλαλήσαντα. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Το μόνο όμως που θέλω να πω είναι ότι είναι πάρα πολύ απογοητευτικό αυτό το σύστημα με το πόσα υγρά μπορεί κανείς να μεταφέρει μαζί του στην καμπίνα του αεροπλάνου. Δεν ξέρω πρόκειται για την πίεση που έχουμε από τα κράτη-μέλη, πρόκειται για την τεχνολογία. Τι είναι αυτό το οποίο μας έκανε να αποτύχουμε και να μην καταφέρουμε να φτάσουμε στο ύψος των φιλοδοξιών μας. Δεν υπάρχει τεχνολογία που να μας επιτρέπει με ασφάλεια να μεταφέρουμε υγρά. Υπάρχει κάποια τεχνολογία που να μπορεί να μας κάνει να διακρίνουμε τα ασφαλή από τα μη ασφαλή υγρά. Αν ναι, πόσο θα κοστίσει μια τέτοια τεχνολογία για να τη χρησιμοποιήσουμε εφόσον υπάρχει. Πολύ θα ήθελα να το ξέρω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνη δεν είναι μόνη στον κόσμο, έχει και τέρους, τρίτες χώρες, από τις οποίες μας έρχονται αεροπλάνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αεροπλάνα έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνε σε άλλες, σε τρίτες χώρες. Ρωτάω λοιπόν, οι εταίροι μας τα ξέρανε, ήταν έτοιμοι να δεχτούν τις δικές μας προδιαγραφές στα δικά τους αεροδρόμια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Φλάκιστάν. Λίγο πολύ λέχθηκαν όλα. Πολύ σύντομα γνωρίζετε κύριε Ρόιτερ ότι είμαι πολύ επιφυλακτικός, ήμουν μάλλον πολύ επιφυλακτικός απέναντι σε αυτό το ενδιάμεσο βήμα αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι χαίρομαι για την έκβαση της υποθέσεως που τη βρίσκω απολύτως απαράδεκτη. Για μένα είναι σημαντικό να πούμε ωστόσο πρώτο δεν κάνουμε άλλα πειράματα, ενδιάμεσα βήματα και το καθεξής που επιβαρύνουν τους επιβάτες εν τέλει. Εμείς βέβαια υποδειγματικοί όπως πάντα έχουμε αγοράσει όλες τις συσκευές και ήμασταν έτοιμοι. Γερμανία δηλαδή. Το 2013 μάλλον ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε θα εξακολουθούν να υπάρχουν. Α μην μπούμε λοιπόν από τώρα ότι δεν και καλά 2013 θα πρέπει να είναι μια ορισμένη δεσμευτική ημερομηνία. Α δούμε ποια πράγματα είναι δυνατόν να γίνουν όπως είπατε το 2012 και ενδεχομένως θα ισχύσει εν τέλει αυτό που είπε η κυρία Φώστερ. Εγώ τώρα η σειρά μου. Πρέπει να ξέρουμε κάτι ξεκάθαρο. Ο κύριος Γκρός ανέφερε τα γεγονότα. Αλλά ας απομακρυνθούμε λίγο από το ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται σε ανησυχίες ασφάλειας. Όχι, για οικονομικούς λόγους. Για οικονομικούς περιορισμούς τα οικονομικά, που δεν μπορούμε να αγοράσουμε τα καινούρια μηχανήματα και όχι το θέμα της ασφάλειας. Εγώ έχω μιλήσει με τους κατασκευαστές και μου λένε τα μηχανήματα τα έχουμε. Μίλησα με τα αεροδρόμια, μου είπαν ότι όχι. Μίλησα με κυβερνήσεις, δεν ξέραν κατά πόσο ήμασταν έτοιμοι ή όχι. Το τελικό όμως ήταν ότι έπρεπε να πληρωθούν τα μηχανήματα αυτά και είναι αλήθεια αυτό που λέει ο κόσμος, ότι δεν είναι το Συμβούλιο που πρέπει να κατηγορήσουμε και εμείς πρέπει να πάρουμε κάποιες ε, ευθύνες που τους επιτρέψαμε να βρούνε διέξοδο. Και αυτό είναι το μάθημα που πρέπει να πάρουμε από αυτή την υπόθεση. Και η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει τις δικές της ευθύνες ότι περίμενε υπερβολικά πολύ μέχρι να φτάσουμε στο παραπέντε και να βρεθούμε αντιμέτωποι με τα προβλήματα. Υπάρχουν και τα λόμπι στα αεροδρόμια και αυτοί δημιουργούν πρόβλημα. Άρα είναι τα λόμπις που δημιούργησαν τα προβλήματα από κοινού με το Συμβούλιο και με όλα τα άλλα που σας είπα πριν και το λέω αυτό ανοιχτά. Αυτή τη θέση θα υποστηρίξουμε όπου και να βρεθούμε. Είναι θέμα κόστους. Τώρα για την ε, ε, ανάμειξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Μα τελικά θα υπάρξουν ε, εμπορικές κυρώσεις εντό εισαγωγικών. Δεν υπάρχουν ε, ανησυχίες ασφάλειας όπως είπαμε, αλλά γιατί οι Αμερικανοί ε, θα διαπιστώσουν ότι έχουν πιο αυστηρά μέτρα τελικά από αυτά που νομίζανε. Και κάτι ακόμα. Για το 2013 Ποιο ξέρουμε, μήπως το 2013 το Συμβούλιο έρθει και πει ακριβώ τα ίδια πράγματα. Αυτό πρέπει να αποφύγουμε. Κάποιος μίλησε για μια δέσμευση, υποχρέωση να αναλάβει το Συμβούλιο. Εσύ το είπες, δημόσια. Μα το Συμβούλιο υπόσχεται ό,τι θέλει και πολύ εύκολα σπάει τις υποσχέσεις του. Εγώ δεν θα καμία εμπιστοσύνη στο Συμβούλιο με τις υποσχέσεις τους. Οι σχέσεις με το Συμβούλιο βρίσκονται σε πολύ κακό επίπεδο ανάμεσα σε μας και το Συμβούλιο. Σήμερα το απόγευμα είχαμε ολόκληρη συζήτηση για μια άλλη υπόθεση για την οποία επίσης το Συμβούλιο δεν τήρησε τις υποχρεώσεις του και τις υποσχέσεις του. Λοιπόν τέτοιες υποσχέσεις από το Συμβούλιο είναι μηδέν. Δεν αξίζουν καν το χαρτί πάνω στο οποίο γράφονται. Οπότε τι κάνουμε. Πρέπει να επιμείνουμε για το 2013. Πρέπει να τα καταφέρουμε το 2013. Δεν θέλουμε δικαιολογίες, δεν θέλουμε ε, να μας πούνε ότι ξέρω εγώ τα λεφτά πήγανε για να σκοτώσουν έναν άλλον ηγέτη της Αλκαΐντα δύο μέρες πριν την ημερομηνία που θέλουμε να εφαρμοστεί το μέτρο. Δεν θέλουμε τέτοια. Έχουμε επιμείνει για το all screening, έχουμε επιμείνει για τα μηχανήματα και αυτό πρέπει να εφαρμοστεί γιατί υπάρχουν τα κράτη-μέλη που δεν το θέλουν ούτε αυτό. Και πρέπει να πετύχουμε συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείε, ώστε να μην είναι αυτοί στο μέλλον που θα μας τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια. και 36 ώρες. Και αυτό είναι ανόητο. Ας ξεχάσουμε τι λέει το Συμβούλιο για αυτά. Αλλά ας προσπαθήσουμε με τις Ηνωμένε Πολιτείες να καταλήξουμε σε μια θέση ώστε να αποφύγουμε για δεύτερη φορά το ίδιο σενάριο. Σαν και αυτό που έχουμε τώρα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Πρέπει να συμφωνήσουμε με αυτά που λέτε. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι μας αφήνει πάρα πολύ πικρή γεύση στο στόμα όλη αυτή η υπόθεση και μπορούν να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν οι συνάδελφοι, αλλά από τις αντιδράσεις που έχω ακούσει εγώ από το Συμβούλιο γι' αυτό και των άλλων, έχουν σαν αποτέλεσμα μια πολύ πικρή γεύση στο δικό μας στόμα της Επιτροπής μας. Για διαδικαστικό κύριε Λεντεμπέργε. Όταν θα απαντήσει ο κύριος Ρόιτερ, μήπω θα μπορούσε να σχολιάσει και το θέμα της τάχτη τώρα του ηφαιστείου. Να μας πει δύο λόγια γι' αυτό. Δηλαδή πάλι για την ε, διαχείριση κινδύνου, καλά. Ο κύριος Ρόιτερ. απαντήστε μας για τα θέματα ασφάλειας και μετά για το σύννεφο στάχτης μας λέτε αν έχουμε ακόμα τους διερμηνείς μαζί μας. Λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ όλα τα μέλη της Επιτροπής αυτής που έδειξαν, ε, δεν θα έλεγα ακριβώ κατανόηση, αλλά εν πάση περιπτώσει η συζήτηση ήταν μετρημένη ε, και βασιζόταν σε αυτά που πραγματικά νιώθετε για αυτή την υπόθεση. Να σχολιάσω κάποια από τα πράγματα που είπατε και θα ξεκινήσω με τον κύριο Τεγράντες. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε ένας βασικός παίκτη στα θέματα ασφάλειας ως Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα υποχωρήσουμε στις τάσεις που υπάρχουν να υπάρχουν ε, εθνικές πολιτικές ασφάλειας από τις χώρες μέλη. Η ρήτρα opt-out στην πραγματικότητα θα ήταν ένας τρόπος, είναι ένας τρόπος επανεθνικοποίησης της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας. Και αν έχετε 25 χώρες μέλη, που χρησιμοποιούν τη ρήτρα opt-out και σας υπενθυμίζω ότι στις διαπραγματεύσεις για τη ρήτρα opt-out της εξαίρεσης κάτι πετύχατε. Και αυτό ήταν ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να αιτιολογήσουν γιατί θέλουν opt-out και η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την αιτιολόγηση αυτή. Αλλά όταν πρέπει να το κάνουμε αυτό για 25 χώρες που ζητούν να χρησιμοποιήσουν τη ρήτρα αυτή opt-out, καταλαβαίνετε πόσο περίπλοκη θα είναι η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουμε για να διαπιστώσουμε τι κάνουν οι χώρες μέλη, αν είναι οικονομικοί οι λόγοι που ζητούν την εξαίρεση ή πραγματικά λόγια ασφάλεια. Και γι' αυτό πριν από τις 29 Απριλίου τι είπαμε, είπαμε εντάξει αυτές οι λίγες χώρες που ζητάνε το opt θα τις πάμε στο δικαστήριο. Αλλά άμα έχουμε 25 είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και υπήρχε και η υπόθεση της Αμερικής. Και αυτό λοιπόν θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι στην πολιτική ασφάλεια εξακολουθούμε να έχουμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Έτσι η γρήγορη αντίδραση και η δικιά σας ε, η άδεια να προχωρήσουμε πιο πέρα και να έχουμε μια γρήγορη αντίδραση που λέει εντάξει μπορεί να μην είμαστε τώρα έτοιμοι είναι ό,τι καλύτερο. Αλλά στη συνέχεια θα είμαστε πιο ισχυροί και θα έχουμε ένα μηχανισμό ο οποίος θα λέει όχι εμπιστοσύνη αλλά έλεγχος. Έρχομαι τώρα στις άλλες παρεμβάσεις. Τα πραγματικά ζητήματα που απέχουν λίγο από αυτό που είπατε εσείς είναι κρατάμε την ημερομηνία 2013 ή το αφήνουμε ανοιχτό για να καταργηθεί ο έλεγχος των υγρών. Θα σας έλεγα λοιπόν, αν θυμόσαστε τα πράγματα όπως και εγώ για τη διαδικασία, η ημερομηνία 2013 είχε ήδη αμφισβητηθεί από το Κοινοβούλιο παλιότερα και γι' αυτό είχαμε και τον διάμεσο αυτό βήμα. 2013 είναι η ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί διεθνώς. Έχετε δηλώσεις των ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστραλίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λένε ότι θέλουμε να σταματήσει αυτό το καθεστώς για τα υγρά το 2013. Προτείνω λοιπόν να μην παραιτηθούμε από την ημερομηνία αυτή. Αλλά, όπως λέει και ο κύριος ε, Κρός, να δώσουμε ένα πραγματικό ραντεβού το 2012 ώστε να εξετάσουμε είναι ρεαλιστική ημερομηνία αυτή του 2013. Υπάρχουν τα μηχανήματα. Τέτοια πράγματα χρειαζόμαστε, αυτό χρειαζόμαστε, γιατί αυτό που πραγματικά θέλουμε και αυτό που θέλετε κι εσείς, να κάνετε τη ζωή των επιβατών πιο εύκολη, ε, δεν θέλουμε να είναι υποχρεωμένοι πια να βγάζουν τα μπουκαλάκια από τις βαλίτσες τους, να έχουν 100 ml μπουκαλάκια και τίποτα άλλο. Πρέπει να είμαστε σε μια διαδικασία. Όπου να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε πού θα βρισκόμαστε το 2012 καταρχήν. Έτσι ώστε να συμμεριστούμε αυτή την προσέγγιση για να υποβοηθήσουμε την κίνηση. Άρα να έχουμε ένα εκούσιο σύστημα κατ' επιλογή, να κρατήσουμε το 2013 και να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να επαναδεσμευτούν για το 2013. Ομάδα εργασίας με τη σύνθεση που είπατε, κράτη-μέλη, η βιομηχανία θα πρέπει επίσης να συμμετάσχει κάπως, με κάποιο τρόπο, να σας δώσουμε πληροφορίες στο Κοινοβούλιο. Επίσης, δέσμευση τον ΗΠΑ για το 2013. Ας εργαστούμε επ' αυτού και δυστυχώς πολλές φορές επανέρχομαι εδώ για να σας πω πώς έχει κατάσταση εν μέσω καθυστερήσεων. Πρόεδρος, δεν ξέρω όμως αυτό το 2013, αυτό το συνονθήλευμα ή μάλλον αυτή η σύναξη του 2013. This committee will meet and oh, it can't be done. Τι νόημα θα έχει το 2012 για να αποφασίσουμε εν ώψη του 2013. Αυτή η σύναξη δεν ξέρω τι νόημα θα έχει για το πού βρισκόμαστε. Δηλαδή αυτή η Επιτροπή 2012 αυτή η επιτροπή ad hoc, α, θα έρθει σε εμά. Και αν εμείς πούμε, α, το 2013 αποφασίσαμε, έτσι και θα έχουν τα πράγματα. Ναι, πράγματι. Τώρα θα προτείνουμε να τροποποιήσετε την υπάρχουσα νομοθεσία, κρατώντας το 2013 με την Επιτροπή Ad Hoc, θα επανέλθουμε το 2012 και θα μας πείτε εσείς ότι ναι, πράγματι έτσι έχουν τα πράγματα, θα τα καταφέρουμε αυτή τη φορά και αυτή την πρόταση θα σας ε, υποβάλω. Άρα κρατάμε το 2013, θα πούμε ότι επί του παρόντος το σύστημα είναι εκούσιο για το 2011 και το 2013 θα αποφανθούμε για τα υγρά με βάση την ομάδα εργασίας που θα έχει συσταθεί και τις ε, συζητήσεις σε διεθνές επίπεδο και τις δηλώσεις που θα έχουμε μέχρι τότε. Εντάχει σας παρακαλώ, γιατί θέλω να δούμε και το ηφαίστειο πριν φύγουν οι διερμηνείς. Θα ήθελα εντάχει να υποβάλω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη έχει ως εξής από όσο γνωρίζετε υπάρχουν σαρωτές υγρών μέχρι τούδε για να ξέρουμε ποια είναι τα ασφαλή και ποια όχι. Α, η απάντηση είναι απλή. Έχουν πιστοποιηθεί μέχρι τώρα, έχουν λάβει πιστοποιητικό δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Civil Aviation Authority πάνω από 10 συσκευές για τον έλεγχο υγρών. Υπάρχουν βεβαίως και διάφορες ποιότητες A, B, C κλπ. Αλλά υπήρχαν αρκετά μηχανήματα διαφόρων κατασκευαστών πριν από τις 29 Απριλίου ε, φέτος στην αγορά. Πρόεδρος, οκ, okay, στάχτη, τέφρα. Ματιέ, αν να ναι, αν... θα μπορούσαμε να μάθουμε και το κόστος των συσκευών αυτών. Για το 2012 θέλω να πω μια λέξη. Όταν πρότεινα κάποια ημερομηνία μέσα στο 2012, θεωρώ ότι οι χώρες μέλη θα πρέπει να γνωρίζουν και ένα έτος πριν ποια πράγματα θα μπορούν και δεν θα μπορούν να εφαρμόσουν. Αυτό που αναμένουμε από το 2012 να μπορούμε να τα συζητήσουμε εδώ στην Επιτροπή Μεταφορών. Να επιστρέψουμε και στα όσα ανέμενε ο κύριος Ελ Χαντράουι πρόσφατα. Δηλαδή μια ξεκάθαρη, ξεκάθαρη θέση του Συμβουλίου, μια ξεκάθαρη θέση της Επιτροπής και μια δηλαδή ξεκάθαρη θέση του Κοινοβουλίου να μπορούμε να πούμε εδώ δηλαδή τι ακριβώς αναμένουμε για το 2012. Τέφρα. Πρόεδρε. Θα πρέπει να μάθουμε μια νέα λέξη. Ε, ε, ε, Το όνομα του ηφαιστείου. του ηφαιστείου στην Ισλανδία. Η κατάσταση τα όλα ξεκίνησαν την, ε, το Σάββατο βράδυ. Την Κυριακή ε, είχαμε έναν πυρήνα ε, σας ανάγκης και με το Eurocontrol προσπαθούμε να δούμε πώς έχει η κατάσταση σε σχέση με τη διάχυση του, της τέφρας. Νομίζω ότι αυτή τη φορά αντιδράσαμε τάχιστα με σπουδή, διότι έχουμε έναν μηχανισμό κατεπίγουσας ανάγκης, ο οποίος ε, ε, συστάθηκε μετά από την ε, κατάσταση του παρελθόντος Απριλίου. Θα υπάρξουν περιορισμοί στις πτήσεις, θα υπάρχουν θέματα ως προς τα δικαιώματα των επιβατών, αυτό είναι σίγουρο, αλλά νομίζω ότι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, δεν έχω βεβαίως την τελευταία ενημέρωση των τελευταίων ωρών, όμως από όσο γνωρίζω δεν είναι η ίδια κατάσταση με την Περσινή, όπου είχαμε πλήρη παράλυση στον μεγαλύτερο τμήμα του εναερίου χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη-μέλη, ακολουθούν μια διαδικασία, τη διαδικασία αυτή που συζητήθηκε και επικυρώθηκε, δηλαδή να έχουμε μία προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο, ανάλυση κινδύνου, για να δούμε κατά πόσο θα πρέπει να εκτελεστεί η πτήση ή όχι και μπορούμε να πούμε ότι τα ηφαίστεια πάντα θα υπάρχουν αλλά τον τελευταίο χρόνο μάθαμε πώς να αντιμετωπίζουμε το ζήτημα αυτό κατά καλύτερο και πιο συντονισμένο τρόπο. Αυτά μπορώ να σας πω επί του παρόντος. Αν μιλήσετε με τους μετεωρολόγους θα σας κάνουν διάφορες προβολές σε σχέση με τη διάχυση του νεφελώματος, τέφρας. Και όλα αυτά τα στοιχεία συνοδεύονται από στοιχεία προειδοποίησης, δηλαδή από όσο γνωρίζουμε, πάντα έτσι αρχίζουν οι μετεωρολόγοι. Αλλά επί του παρόντος ε, αποδεικνύουμε και δείχνουμε ότι μπορούμε να συντονίζουμε καλύτερα τα πράγματα από την τελευταία φορά. Υπάρχει ε, η μονάδα κρίσης τα κράτη-μέλη συντονίζουν μεταξύ τους. Ο Αντιπρόεδρος Κάλλας ήρθε σε επαφή με την Ουγγρική Προεδρία, συζήτησε και με τους υπουργούς η χώρα των οποίων πλήττεται ιδιαίτερα και ούτω καθεξής. Θα συνεχίσουμε στα αγγλικά έτσι ώστε οι διερμηνείς να μπορέσουν να αποχωρήσουν. Oh, uh,